Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίασή μας. Για οικογενειακού λόγου, η κυρία Παλιαδέλη ζήτησε να μην παρουσιάσει την έκθεσή τη σήμερα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρέπει να αναβληθεί αυτό για οικογενειακού λόγου. Και κατά την επόμενη συνεδρίαση στις 23 και 24 Ιουνίου θα συζητήσουμε το σχετικό θέμα. Όμω, όμως στις 28 θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Ähm, και έτσι λοιπόν προτείνω ένα σημαντικό θέμα να ξεκινήσουμε, ένα σημαντικό θέμα ποδόσφαιρο UEFA και δεν είναι μόνο θέμα γερμανικό από ό,τι φαίνεται αλλά και των περισσότερων άλλων χωρών. Αλλά το ξέρω ακριβώς διότι στην οικογένειά μου υπάρχουν τόσοι τρελοί φανατικοί ποδοσφαιρόφελοι που δεν ξέρω πού να καταφύγω για να γλιτώσω μια τέτοια αναμετάδοση. Λοιπόν, θα έρθουμε αμέσως αυτό. Τώρα, όπως έχει η ημερήσια διάταξη και τροποποιήθηκε, εγκρίνεται, δεν υπάρχουν ενστάσεις, περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Θα έχετε τα πρακτικά μπροστά σας. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αξιολογήσετε. Αν μέχρι του τέλους της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις, τότε θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται συνολικά τα πρακτικά αυτά. Περνάμε στο σημείο 3 τη ημερήσιας διάταξη, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Να σας πω μόνο δεν υπάρχουν ε, σουηδικά, εσθονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, για κάποιες γλώσσες ε, οι Ολλανδοί μπορούν να ε, μιλήσουν. γερμανικά όμως δεν θα υπάρχει διερμηνία αντίστοιχη. Λοιπόν, συγγνώμη. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Χαιρετίζω τον κύριο Γκαγιά και τον κύριο Τραβέσο. Πρωτού δώσω τον λόγο σε εσά, θα ήθελα να πω γιατί σας προσκαλέσαμε κύριοι. Σας χαιρετίζω θερμά και ξέρω ότι ο κύριος Γκαλιάχου είναι και σύμβουλος του κυρίου Πλατινή και ο κύριος Τραβέσο είναι ο επικεφαλής της αδειοδότησης ε, ποδοσφαιρικών ομάδων ηλεσχών. Σημαντικά θέματα αυτά και προσωπικότητες. Παρακαλέσαμε να έρθετε σε εμά για να μας πείτε ποιοι είναι οι νέοι οικονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν ακριβώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα αντιδρούμε εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είμαστε πάντα πάνω-πάνω και πάντα πανέτοιμοι. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για αυτό το θέμα έχουμε ήδη αρκετέ φορέ ασχοληθεί με αυτό. Πολλέ υπερβολικά πολλέ λέσχε έχουν μεγάλα ε, ελλείμματα και χρέη και έχουν ε, ανοίξει τέτοια χρέη ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν τη δυνατότητά τους για αγορά παικτών. Και υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις, πολύ ακραίες περιπτώσεις, που έχουν και θλιβερό τέλος. Όλο αυτό είναι κακή εικόνα των, των ποδοσφαιρικών λεσχών και δεν είναι και ανταγωνισμός, δεν είναι πραγματικός ανταγωνισμός. Όπως και στην χρηματοοικονομική κρίση το ζήσαμε, υπάρχουν πολλές φούσκες, ε, σκάνε αυτές ε, και έτσι κρίμα για όσους εμπλέκονται σε αυτές τις λέσχες ε, και υφίστανται τις συνέπειες. Χαιρόμαστε για το ότι προβληματίστηκε η UEFA να δει τι μπορεί να γίνει και κατέληξε και σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι, και αυτό πάντα το έλεγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερο εύρο ανταγωνισμού. Ένα πιο ισόρροπο ανταγωνισμό στι ομαδικέ στα ομαδικά παιχνίδια. Όχι μόνο σε αυτό το ποδόσφαιρο και σε άλλα ομαδικά παιχνίδια. Γι' αυτό αδειμονούμε να ακούσουμε τι σκέφτηκε να κάνει η UEFA και τι προτείνει και αν πιστεύει ότι όλα αυτά θα είναι αποτελεσματικά και με ποιο τρόπο οι κυρώσει θα λειτουργούν και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Να σας πω ότι έχουμε μία ώρα για αυτό το σημείο συνολικά και θα ήθελα <clears throat> για τη συζήτηση να το αναφέρω αυτό. Ξεκινάμε. Οι δύο κύριοι θα έχουν τον λόγο. Μπορείτε να συμφωνήσετε ποιος θα ομιλήσει πρώτος. Θα δίνω την δυνατότητα αυτά τα οποία αποφασίσατε να μας τα παρουσιάσετε με ε, κατανοητή, εύληπτη γλώσσα. Παρακαλώ, εσύ έχει τον λόγο. Εσείς κύριε Γάγια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης που μας ε, κάλεσε να μιλήσουμε για τα οικονομικά θέματα. Είναι πολύ φυσιολογικό το έγγραφο αυτό το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δοθεί εμάς πρώτα. Γιατί η πρωτοβουλία του οικονομικού fair play και των οικονομικών κανόνων της άδεια. Ε, η πρωτοβουλία λοιπόν προέρχεται από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την προηγούμενη μάλιστα νομοθετική κοινοβουλευτική θητεία και πιο συγκεκριμένα την έκθεση Μπέλετ και την έκθεση Μαυρομάτη για την Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αθλήματα. Με βάση αυτές τις δύο εκθέσεις, πολύ σύντομα, πολύ νωρίς, υποδείξαμε το οικονομικό πρόβλημα, τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ειδικά οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Και μας ζήτησαν να εργαστούμε ε, σε επίπεδο αδειών για να υπάρχει οικονομική σταθερότητα, οικονομική διαφάνεια και ισορροπία στους, στα διάφορα γεγονότα, ε, πλαισιώνοντας αυτό το σύστημα διών. Στις αρχές του 2009 αρχίσαμε να δουλεύουμε, διορίσαμε μία ανεξάρτητη επιτροπή ε, ελέγχου των οικονομικών των ποδοσφαιρικών ομάδων υπό την προεδρία ενός συναδέλφου σας του Jean-Luc Deanna και με αυτή την πρωτοβουλία ε, την ίδια στιγμή που ξέσπαζε η παγκόσμια οικονομική κρίση, εμείς στρεφόμασταν σε αυτά τα θέματα τα οικονομικά. Ε, αυτή η σύμπτωση δείχνει και τα προβλήματα τα οποία οι ευρωπαϊκές ε, ποδοσφαιρικές ομάδες αντιμετωπίζουν. Και βεβαίως ε, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιτάθηκαν λόγω της κρίσης. Οι δύο εκθέσεις Μπελέτ και Μαυρομάτι τονίζουν ότι υπάρχει χρέωση, όλο ένα και μεγαλύτερη χρέωση λόγω των μισθών που πληρώνουν στους παίχτες. Την, ε, την περασμένη εβδομάδα, μετά από συζητήσεις που δίρκεσαν περίπου εννέα μήνες και με μια πολύ ενδελεχή διαβούλευση με τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τους παίκτες, τις ομοσπονδίες και την ε, Ένωση, προωθήσαμε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποιους κανόνες για οικονομικό και η ισοτιμία, fair play, για να ενδυναμωθεί το σύστημα των αδειών. Και μαζί με τον συνάδελφο, ε, θα δώσω μάλλον τον ε, λόγο στον συνάδελφο τώρα, ε, τον κύριο Τραβέσο, ο οποίος θα σας κάνει μια παρουσίαση πολύ πιο τεχνική από αυτή που ακούσατε μέχρι στιγμή. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, Μεγάλη τιμή κάνατε στην ε, UEFA που μας προσκαλέσατε, που μας προσκαλέσατε εσείς και η κυρία Πακ. Ε, για να σας παρουσιάσω τις ε, βασικές αρχές της ε, μεταρρύθμισης που μόλις προώθησε η Επιτροπή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια μεταρρύθμιση που θέλησε ο πρόεδρος Πλατινή, ο οποίος άκουσε την, το καμπανάκι που προέρχεται από τις ποδοσφαιρικές ομάδες, από τους επαγγελματίες προς την UEFA. Τα τελευταία χρόνια ε, επλήγησαν όλα τα σπορ και ιδιαίτερο το ποδόσφαιρο. Οι πρόσφατες αποτυχίες και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, πάρα πολλές κοινωνίες σε πολλές χώρες ε, είναι η απτή και δυσάρεστη μαρτυρία. Μία μεταρρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Γκαγιά, θα γίνει πολύ σύντομα, λόγω του κατεπήγοντος του θέματα, με την ε, υποστήριξη όλων των διαφερομένων και με την ε, συνεργασία πολλών εμπειρογνωμών του κλάδου. Πριν σας παρουσιάσω τα πιο περίπλοκα θέματα του οικονομικού fair play, θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η UEFA έβαλε τις βάσεις αυτής της μεταρρύθμισης ήδη με την εισαγωγή του 2004 του συστήματος των ε, αδειών UEFA. Ένα σύστημα που βασίζεται σε ελάχιστα πρότυπα και ε, αρχές καλής ε, διαχείρισης που πρέπει να σέβονται όλες οι ομάδες, ούτω ώστε να μπαίνουν στις διεθνείς, στα διεθνή συμβάντα, στις διεθνείς διοργανώσεις που διοργανώνει η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες ε, είχε πει ότι το σύστημα αδειών δεν προβλέπει απλώς οικονομικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια σε άλλους τομείς. Φερρυπίν προβλέπει ε, αθλητικά κριτήρια, όπως η κατάρτιση των, ε, και εκπαίδευση των νέων, ε, αθλητική εκπαίδευση και παιδεία, αλλά και αντιντόπι, ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού, επίσης διοικητικά κριτήρια, ούτω ώστε στο εσωτερικό των ποδοσφαιρικών ομάδων να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα, τις κατάλληλες δεξιότητες, ούτω ώστε να βελτιώσουμε ε, την ασφάλεια και την ποιότητα των εγκαταστάσεων. Επίσης, οικονομικά κριτήρια, αυτά είναι μια ολόκληρη δέσμη. Τα τελευταία χρόνια χάρη σε αυτά αυξήσαμε τη διαφάνεια, την οικονομική διαφάνεια και μέσω των ελέγχων που κάνει η UEFA προστατεύουμε την ακαιρεότητα και την καλή διεξαγωγή των διοργανώσεων. Το σύστημα των αδειών ε, εισήχθη και στις 53 ε, ομοσπονδίας μέλη της ΣΟΕΦΑ. Σε 45 από αυτές υιοθετήθηκε ως αρχή καλής διαχείρισης και σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση στις, ε, στις εσωτερικές διοργανώσεις, εθνικές διοργανώσεις. Μιλάμε για 800 άτομα χωρί να μιλάμε για αυτού που ασχολούνται στο επίπεδο παιδοσφαιρικών ομάδων. Κάθε χρόνο πάνω από 600 άτομα ζητούν μια άδεια UEFA για να έχουν πρόσβαση στι διεθνεί διοργανώσει και σε ό,τι αφορά τι δικέ μα διοργανώσει, τα τελευταία χρόνια 49 ομάδε ε, δεν έγιναν δεχτές στις διοργανώσεις UEFA γιατί δεν είχαν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ε, τα ελάχιστα πρότυπα και στάνταρ. Το σύστημα των αδειών δεν επέτρεψε και ούτε ήταν καν ο στόχος τον περιορισμό των στόχων, τον περιορισμό των δαπανών σε ό,τι αφορά τα κόστη για τους ποδοσφαιριστές και, και τη μεταφορά από τόπο σε τόπο. Με βάση μια μελέτη που έκανε πρόσφατα η UEFA, Φαντάζομαι ότι έχει μοιραστεί εδώ στην αίθουσα, γιατί είχαμε προβλέψει διάφορα αντίτυπα εδώ και υπάρχουν στην αίθουσα τα συσσωρευμένα, οι συσσωρευμένες απώλειες το 2008 όλων των ομάδων ε, της πρώτης κατηγορίας ε, είναι 58 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Γιατί δώστηκαν, δόθηκαν ε, πριν και μισθή σε ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ψηλή. Σε ορισμένε χώρε έχουμε ακόμα ψηλότερους μισθούς ε, και σε 57 ποδοσφαιρικές ομάδες έχουμε πραγματικές ε, υπερβάσεις. το 35% των ποδοσφαιρικών ομάδων έχει ε, αρνητικό ίδιο κεφάλαιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το χρέος, αυτό αυξάνεται. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας το χρέος ε, απέναντι στα πιστοτικά ιδρύματα, φτάνει στα 5,5 ε, δις μόνο το 2008. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, μακροπρόθεσμα. Και με βάση μια ανάλυση που κάναμε, δεν νομίζω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και μάλιστα ε, ήδη είδαμε ότι το 2009 η κατάσταση χειροτέρεψε και σε αρχέ του 2010 έτσι περαιτέρω. Εξού και η πρωτοβουλία του οικονομικού fair play. Το 2009, όπω εξήγησε ο Γιάνν Φίγκελ, πρώην Επίτροπο ε, Εκπαίδευση και Αθλητισμού, τα νέα μέτρα του οικονομικού fair play πρέπει να συμπληρώσουν το σύστημα των ε, αδειών που υπάρχουν ήδη ο νέος κανονισμός τώρα που θα είναι στη διάθεσή σας ε, στο ιστοσελίδα της UEFA έχει κριτήρια για την εκχώρηση αδειών και νέες ε, προϋποθέσεις για το οικονομικό θεραπεία. Όλα αυτό, όλοι αυτοί οι κανόνες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, τους ποδοσφαιριστές, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ακόμη και τους ε, φιλάθλους μία διαδικασία διαβούλευσης που κράτησε περίπου ένα χρόνο και που ενεπλάκησαν εργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και νομίζω ότι το στόχο όλοι το συμμεριζόταν. Ε, εκπονήθηκαν μάλιστα και κανόνες με πάρα πολύ λεπτομέρειες τεχνικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ε, θέλουν να υλοποιηθούν οι εξή στόχοι. Να βελτιωθεί η οικονομική ικανότητα των ποδοσφαιρικών ομάδων, αυξάνοντα την διαφάνεια και την αξιοπιστία. Να εξασφαλίσουμε ότι οι ποδοσφαιρικέ ομάδε ε, αναλαμβάνουν τι ευθύνε και τα χρέη του απέναντι στου υπαλλήλου, στου παίχτε, ε, στα, στις κοινωνικές και και οικονομικού ε, θεσμούς μέσα στι ε, προθεσμίε που προβλέπονται. Μεγαλύτερη προθεσμία και οικονομικό ορθολογισμό ε, στο ποδόσφαιρο σε όλε τι ομάδε Να, να προστατευτεί η ακαιρεότητα και η καλή διεξαγωγή των διοργανώσεων και να ενθαρρύνουμε τι ποδοσφαιρικέ ομάδε να περιορίσουν τι δαπάνε και να προωθήσουν τις επενδύσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν μακροπρόθεσμα κέρδη. Και επομένως να προστατευτεί η η δυνατότητα να παραχθούν μακροπρόθεσμα κέρδη ε, και να υπάρξει βιωσιμότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι στόχοι αυτοί λένε ότι η UEFA έχει το καθήκον να διασφαλίσει το περιβάλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μέσα στο οποίο ανταγωνίζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Να μειωθεί αυτή η πληθωριστική τάση των ποδοσφαιρικών ομάδων που έχουν μια τάση να δίνουν όλο και μεγαλύτερους μισθούς, κυρίως τους παίχτες. Ε, και ε, κατά τις μεταγραφές. Ε, το slide αυτό δείχνει ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις του οικονομικού fair play και πώς εντάσσονται με, τα, το σύστημα των αδειών. Από κοινού θα μας επιτρέψουν να, έχουμε, να υλοποιήσουμε τους στόχους και θα αναλάβουμε υπόψη μας όλα τα οικονομικά στοιχεία. Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ κερδών και και εξόδων, ε, ρευστότητα. Τα, οι ποδοσφαιρικές ομάδες θα πρέπει να ζητήσουν μία άδεια, να σέβονται τα κριτήρια των αδειών που έχουν ε, δημιουργηθεί, ούτω ώστε να υπάρχει ε, αξιοπιστία οικονομική βραχυπρόθεσμα. Οι ομοσπονδίε δίνουν τι ε, άδειε για να συμμετάσχει κανεί στι διεθνεί διοργανώσει και αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομάδα πήρε την άδεια και έχει να, να συμμετάσχει στι διοργανώσει μα. Θα μπει σε μια φάση παρακολούθηση, monitoring, αξιολόγησης πολυετούς με σκοπό να έχουμε μία πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση ε, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εν γέννη. Σε αυτή τη φάση της παρακολούθησης θα ζητήσουμε από μια Οικονομική Επιτροπή Ελέγχου των Ποδοσφαιρικών Ομάδων υπό την προεδρία του συναδέλφου σας του Ζαν Λουκ Ντεάν, ο οποίος δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα στην ε, συνεδρίαση για να σας μιλήσει ε, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αυτό το monitoring θα βασιστεί στο, στον κίνδυνο, ούτω ώστε να ελέγξουμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες που δείχνουν δείγματα ανησυχητικά. Θα κάνουμε μία αξιολόγηση και η Επιτροπή αυτή Οικονομικού Ελέγχου θα λάβει υπόψη όλα τα κριτήρια εξατομικευμένα, αλλά και συνολικά τα κριτήρια αυτά θα τα αντιμετωπίσει μέσα σε ένα πλαίσιο δηλαδή. Θα δούμε. Ε, Παραδείγματο χάρη, μπορεί να θεωρηθεί μια συμπεριφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα ε, ω αποδεκτή, αλλά μπορεί να θεωρηθεί η συγκεκριμένη ίδια συμπεριφορά απαράδεκτη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εν γέννη. Μια νέα, ε, μια νέα προϋπόθεση επίσης είναι ο εξοσκελισμός, ο ισοσκελισμός, συγγνώμη, του, του ισολογισμού των ποδοσφαιρικών ομάδων. Και ενθαρρύνονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες να φτάσουν σε ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα. Σε όλες, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν πάρει την άδεια από την Ομοσπονδία τους, απαιτείται αυτό, αυτή η προϋπόθεση και που συμμετέχουν σε διοργανώσεις του, της UEFA. Επομένως, μία ποδοσφαιρική ομάδα πάντα θα πρέπει να ισοσκελίσει τον ε, ισολογισμό της. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι πολύ περίπλοκο, πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Ε, γι' αυτό δεν θα κάνουμε μία αξιολόγηση ετήσια βάση, αλλά μια μεσοπρόθεσμη, πολυετή αξιολόγηση. Μιλάμε για μία τριετή περίοδο αναφοράς πιο συγκεκριμένα. Σε περίπτωση που σε αυτή την περίοδο αναφοράς ε, τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, τότε η ποδοσφαιρική ομάδα θα θεωρηθεί ότι σέβεται την προϋπόθεση εφόσον το μείον της αυτό καλύπτεται από συνισφορές από αύξηση του κεφαλαίου, ε, δωρεές από τους μετόχους της. Ε, οι συνεισφορές υπομορφή δανείου δεν θα ληφθούν υπόψη για να θεωρηθεί ότι η ομάδα πληρεί το κριτήριο. Για την παρέκκληση την αποδεκτή, αυτό προβλέπεται μέσα σε, για 45 εκατομμύρια ε, σε μια τριετία για τα τρία πρώτα χρόνια, δηλαδή 15 ε, εκατομμύρια το χρόνο μπορεί να έχουμε ε, έλλειμμα και θα πρέπει τα επόμενα τρία χρόνια να κατέβει στα 30 ε, εκατομμύρια. Δηλαδή να φτάσει σε ένα μέσο όρο 10 εκατομμύρια το χρόνο το έλλειμμα. Επίσης, πρέπει να υπενθυμίσουμε σε περίπτωση που τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα και η διαφορά οφείλεται σε σε επενδύσεις που γίνονται μακροπρόθεσμα, παραδείγματο χάρη επενδύσεις σε υποδομές. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι δαπάνες που συνδέονται με επενδύσεις ε, σε εγκαταστάσεις, σε στάδια, ε, καταστάσεις προπόνησης κτλ. Ή επενδύσεις για να βγουν νέα ταλέντα ή έξοδα για κοινωνικά προγράμματα, προγράμματα σε διάφορες κοινότητες και κοινωνικές ομάδες, αποκλείονται από το λογαριασμό και δεν λαμβάνονται υπόψη σε ό,τι αφορά την απέτηση για ισοσκελισμό του ισολογισμού. Βεβαίως θα αξιολογούνται πάντα οι ποδοσφαιρικές ομάδες με βάση την ρευστότητά τους, γιατί θα πρέπει πάντα να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους και τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν ως επιχείρηση. Πέρα από τον κανόνα αυτό για τον ισοσκελισμό υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που έχουν εισαχθεί και έχουν υπογραμμιστεί. Παραδείγματος χάρη, να μην υπάρχουν χρέη παλιά, ούτω ώστε να μπορεί η εταιρεία να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους υπαλλήλους, στα, στα πιστοτικά ιδρύματα, ε, κατά τη διάρκεια όλων των διοργανώσεων, ούτω ώστε να μην έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες που συμμετέχουν ε, στις διοργανώσεις μας και που παράλληλα ε, οφείλουν ποσά ε, σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες που συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση. Επίσης, οι ποδοσφαιρικές ομάδες θα πρέπει να στέλνουν μία σειρά από έγγραφα προσωρινά για τον προϋπολογισμό, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουν απαραίτητους πόρους, απαραίτητη ρευστότητα, ούτως ώστε να αναλάβουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τελικά τον, το, την προϋπόθεση για ισοσκελισμό του ισολογισμού τα επόμενα χρόνια. Επομένως, τα μέσα και οι στόχοι του οικονομικού fair play έχουν σαν σκοπό να περιοριστούν, να συμπιεστούν ε, οι δαπάνε, να λειτουργήσουν καλύτερα οι εταιρείε, ούτω ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα. Πρόκειται για μία προσέγγιση που σκοπό έχουμε να βελτιώσουμε τα στάνταρ και όχι μία προσέγγιση με σκοπό να επιβάλλουμε κυρώσεις και να τιμωρήσουμε. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να εφαρμόσουμε κυρώσεις, το σύστημα προβλέπει μέσω φάσεων συνεχών παρακολουθήσεων πολυετών να παρεμβαίνουμε με τρόπο στόχοθετημένο, προοδευτικό και αναλογικό με βάση το, τη σημασία της παράβασης. Πέρα από τη εισαγωγή των νέων ε, κανόνων, θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα στις ποδοσφαιρικές ομάδες να προσαρμόσουν τις δομές τους, τις νέες προϋποθέσεις. Επομένως, από την επόμενη χρονιά, το 2011, οι πρώτες προϋποθέσεις για την έλλειψη παλιών χρεών και την ε, υποχρέωση αποστολής ε, προσωρινών πληροφοριών και από το 2012 θα ακολουθήσουν ε, οι προϋποθέσεις για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού. Θα επιβληθεί δηλαδή και αυτή η αυτό το στάνταρ. Όπως είπε και η Επίτροπος Βασιλείου, αυτή η πρωτοβουλία της ΣΟΕΦΑ είναι πολύ θετική. Έγινε θετικά δεκτή από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι μεταφράζει σε συγκεκριμένα έργα ε, τη σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα ε, προκαλέσει, θα επιφέρει μάλλον σταθερότητα, βιωσιμότητα και θα ανθίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο χάρη σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν θα πρέπει να πληρώνει κανείς περισσότερα από όσα εισπράττει. Είναι πολύ απλή συμπεριφορά αυτή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το συζητάει κανείς αυτό επί ώρες, εφόσον δεν τηρείται τον απλό κανόνα αυτό. Αυτό ισχύει πάνω, δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο και η οικονομική κρίση σχετίζεται με αυτό. Έτσι ξαναφτάνουμε στο θέμα που γενικά μας απασχολεί, ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας ε, και το ίδιο κάνουν και οι ποδοσφαιρικές λέσχες. Αλλά και οι δύο σας ε, αποφύγατε ένα θέμα. Τι γίνεται με τις κυρώσεις, υπάρχουν κυρώσεις. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Μπορείτε να την απαντήσετε μετά όταν απαντήσετε και στου άλλου ε, συναδέλφου. Ο συνάδελφος Μπέλετ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, Ήβο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ντόρι. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους τη ΟΕΦΑ που ήρθαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι αυτά που προτείνονται είναι πολύ σημαντικό βήμα, ε, πολύ καλή εξέλιξη. Υπάρχουν διάφοροι στόχοι. Η ε, ενίσχυση της ισορροπίας, ε, η ενίσχυση της, ε, του ανταγωνισμού είναι θέματα που έχουμε τονίσει σε εκθέσεις μας το 2006 και το 2007 που υιοθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, αυτά αναφέρει ο κύριος Γκαγιά. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα μέτρα που προτείνετε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις, κυρία Πακ. Καταρχήν, έχω την ίδια ερώτηση με εσάς. Ε, τι γίνεται με τις κυρώσεις. Δεύτερον, ελπίζω ότι τα πολλά παραθυράκια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, οι λέσχες, ε, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, δηλαδή για να αποφύγουν τα προβλήματα, θα κλείσουν. Και μία παρατήρηση που σχετίζεται άμεσα με το θέμα αυτό της οικονομικής δικαιοσύνης, του οικονομικού fair play. Όταν μιλάμε για την ανταγωνιστική ισορροπία στους ε, ευρωπαϊκούς ε, αγώνες ε, στο, στον επαγγελματικό αθλητισμό. Νομίζω ότι ο, ήδη ο πρόεδρος Πλατινή της UEFA έχει σημειώσει σημαντικές προόδους για να πετύχει καλύτερη ανταγωνιστική ισορροπία στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Θα πρέπει όμως να ακολουθήσουμε πιο πέρα το δρόμο αυτό για να έχουμε καλύτερη ανακατανομή του πλούτου των χρηματικών πόρων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και μιλάμε φυσικά και για τηλεοπτικά δικαιώματα. Όπως σας είπα, ο κύριος Πλατινίδη έχει σημειώσει ε, σημαντική πρόοδο, αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε περαιτέρω την κατεύθυνση αυτή για να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες ομάδες ε, από τη μία και τους μεγάλους αγώνες ε, και τις ε, μικρότερες ομάδες και τους λιγότερο σημαντικούς αγώνες από την άλλη μεριά. Είμαστε πεπισμένοι ότι όλα τα μέλη της UEFA θα πρέπει να ακολουθήσουν τη μέθοδο της συλλογικής πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει σε, πολλές, σε πολλά μέλη της UEFA, όχι όμως σε όλα. Και πιστεύω ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος ε, και προς αυτή την κατεύθυνση. Και μία τελευταία παρατήρηση, κυρία Πακ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην επόμενη μας πρωτοβουλία, την επόμενη πρωτοβουλία που θα έπρεπε να αναλάβει το Κοινοβούλιο, που έχει να κάνει με τους μάνετζερ των παικτών. Έχουμε ετοιμάσει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη σύνοδο. Έχουμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο ψηφίσματο και αυτό το θέμα σχετίζεται με την δικαιοσύνη στου διεθνεί αγώνε. Προτείνουμε και ελπίζω η UEFA να συμφωνεί να επιμείνουμε οι μάνετζερ των παικτών να μην μπορούν να Ε, εισπράττουν αμοιβή όταν ε, οργανώνεται η μεταγραφή παικτών ε, κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που προτείνουμε και αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση της δικαιοσύνης στους διεθνείς αγώνες. Ε, συνοψίζοντας, κυρία Πακ, ελπίζω ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εργασίας και ότι δεν αποτελούν την τελευταία φάση της ΟΕΦΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις καινοτομίε που έχετε βάλει, για το οικονομικό fair play και για τους κανόνες για τις άδειες στα, για τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ιδίως υπάρχει ε, ένα πρόγραμμα για να εκπαιδευτούν οι νέοι για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Χαίρομαι για αυτό το πρόγραμμα. Ποια είναι η θέση της ΣΟΕΦΑ για τις μεγάλες ξένες επενδύσεις, αραβικές ε, ή ασιατικές, που αγοράζουν ε, ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες. Πιστεύετε ότι μπορούν, μπορούν τέτοιες εξαγορές να δημιουργήσουν ε, μετά τις αρχικές, τα αρχικά ωφέλη προβλήματα, μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Έφτασα με καθυστέρηση, δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την παρουσίαση. Θα ήθελα όμω δύο σχόλια να κάνω. Πρώτο, ότι εγώ πιστεύω ότι πέρα από τις κυρώσεις, το τμήμα των πέρα από πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι μεγάλες λέσχες ότι πρέπει να προσαρμόσουν πώς να το πω, τα είσοδά τους και τα χρέη τους, τις δαπάνες τους. Ένα σύστημα κυρώσεων δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό πιστεύω. Πιστεύω περισσότερο στο να πείσουμε τις λέσχες να δράσουν σωστά και κάνοντας ε, λόγο για τα τηλεοπτικά φοβούμε ότι σε σχέση με τις ε, ισπανικές λέσχες ε, για τα δικαιώματα τους που άμεσα θα είχαν θα έπρεπε να πιστεύει κανείς ότι θα είναι δύσκολο να αποπέμψουν αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Μισή Χάνιμπαλ. Χάνιμπαλ παρακαλώ. Όχι. Δεν θέλετε να παρέμβετε. Ο κύριος Μπόρις παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θα ήθελα να ακούσω από τους εκπροσώπους, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της ΣΟΕΦΑ για την μεταρρύθμιση αυτή. Αυτή η μεταρρύθμιση γίνεται σε μια καλή χρονική στιγμή, διότι αυτά που αφορούν την υπερχρέωση των μεγαλύτερων ομάδων, των μεγαλύτερων λεσχών και αυτό που έχει συμβεί μέχρι στιγμής, θα έχει οδηγεί σε μια μη ε, σχέση όσον αφορά την χρηματοοικονομική υποστήριξη. Η επιτυχία είναι σημαντική φυσικά, αλλά το σύστημα fair play, το ε, δίκαιο παιχνίδι, είναι ένα από τα κυριότερα μέσα για να καταφέρουμε σε σχέση με τις τιμές ε, να ε, σημειώσουμε κάποια μείωση. Πρέπει να είναι λογικές οι τιμές, να μειωθούν, να είναι πιο προσιτές. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και κάτι, το οποίο μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό, να κάνω μια ερώτηση σχετικά. Πρόκειται εδώ για πώς να το πω, για την αναθεώρηση των οικονομικών των ομάδων που αντιμετωπίζουν κινδύνους. Βλέπετε να συμβαίνει ένα τέτοιο monitoring, μια τέτοια επιτήρηση ή εποπτεία που θα επεκτείνεται και σε ομάδες, πώς να το πω, νεότερων ποδοσφαιριστών ή νέων ποδοσφαιριστών της επόμενης γενεάς. Είναι δύσκολο αυτό ίσως σε σχέση με τα τεταμένα οικονομικά των ομάδων. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια τέτοια, ένας τέτοιος συντονισμός, να επενδύουμε στις νεότερες γενιές. Καμιά φορά και συχνά δαπανούμε τεράστια ποσά για παίκτες που προέρχονται από την Αφρική, την Νότια Αμερική. Το σύστημα χρηματοδότησης και της ε, ρύθμισης των χρεών δεν λειτουργεί στην Ευρώπη όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν κάνουμε λόγο για τις οικονομικές πτυχές. Μαρία. Ευχαριστώ. Μαρία Μπαδία Κουτσέτ παρακαλώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ίδια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της UEFA για την εισήγησή τους, τις παρουσιάσεις τους, για αυτή την πρόταση του fair play, του δίκαιου οικονομικού παιχνιδιού. Και προφανώς αυτά τα οποία προτείνονται είναι θέματα που διέπονται από τον κοινή λογική, από τον κοινό νου και είναι σκόπιμες προτάσεις. Ερώτηση για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Και κάπως σε σχέση με το εσείς ίσως προβλέπετε ποια θα είναι και τα προβλήματα ίσως όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια. Ποια προβλήματα μπορείτε να δείτε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αν σκεφτήκατε επίσης για το πώς θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα που θα αναφύονται. Ευχαριστώ. Και τώρα στον τελευταίο γύρο η κυρία Herbert και μετά μπορείτε να δώσετε τις απαντήσεις. Θα έρθουν οι επόμενοι τέσσερις μετά. Παρακαλώ εσείς κυρία. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτού του νέου συστήματος κύριε. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό ως ε, αφετηρία, ως προσέγγιση αυτό το σύστημα να μπορέσει να θέσει σε τάξη τα πράγματα των ομάδων. Και εγώ διαρωτήθηκα γιατί πήρε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα Κάτι το οποίο είναι σχετικά αυτονόητο για αυτονόητα πράγματα τα οποία έπρεπε να λειτουργήσουν. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι ότι υπάρχουν αυτέ οι προτάσει. Τώρα, δύο ερωτήσει. Πρώτον, και εγώ σκέφτηκα μέσω στο θέμα για τι κυρώσει. Κάτι θα μα πείτε σίγουρα για το θέμα των κυρώσεων και αδειμονώ να ακούσω τι θα μα πείτε. Το δεύτερο θέμα, αυτά τα οποία εκπονήσατε θα ισχύουν καταρχήν για ομάδε που συμμετέχουν ε, στο πρωτάθλημα της UEFA μέσα σε τέτοιες συναντήσεις αθλητικές. Έχετε σκεφτεί αυτές οι ομάδες ε, να, ε, να μπορέσει αυτό το σύστημα αδειοδοτήσεων να ισχύσει και για περαιτέρω ομάδες. Διότι αυτό θα ήταν θετικό αν όλες οι εθνικές ομάδες θα μπορούσαν σε σχέση με αυτό το σύστημα να εντάσσονται σε αυτό. Σημαντικό πάντα είναι πιστεύω εγώ το θέμα της προώθησης των νέων ποδοσφαιριστών, της νέας γενιάς. Είπατε ότι σε σχέση με τα κοινωνικά, οικονομικά ε, και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και για τη νέα γενιά, λαμβάνονται αυτά υπόψη στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που έχουν οι ομάδες. Όμως αυτό και πάλι είναι μια προσέγγιση για να μπορέσει κανείς να υπολογίσει τι θα γίνεται τελικά και μήπως δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στο τέλος τέλος οι κυρώσεις. Μήπως κάτι θα πρέπει να γίνει περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, για να μην έχουμε μόνο μια επίφαση αλλά και αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Καγιά θέλετε να λάβετε τον λόγο γι' αυτό, να απαντήσετε. Okay. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Euh, ο, τραβε... ο κ. Τραβέρσο θα μιλήσει για τις κυρώσεις. Και συνεχεία εγώ θα μιλήσω για τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ. Για τις κυρώσεις προβλέπονται και θα εφαρμόζονται προοδευτικά. Οι ομάδες θα παρακολουθούνται μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα τριετίας. Αν την πρώτη χρονιά έχουν ε, προβλήματα, θα λάβουν μια κοινοποίηση και μια προειδοποίηση. Τη δεύτερη χρονιά μπορεί να τους επιβληθούν ε, χρηματικές κυρώσεις. Ε, μπορεί ένα τμήμα των συνεισφορών που προέρχονται από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να τις κρατήσουμε ε, και μπορεί να τους, ε, μπορούν κυρίως αυτές να φτάσουν μέχρι και τον αποκλεισμό από τις διοργανώσεις. Φυσικά όλα εξαρτώνται από την σοβαρότητα της παράβασης, από την τάση που δείχνει η ομάδα. Αν έχει γενικές ε, τάσεις, είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά μας από ό,τι αν έχει αρνητικές. Για τα παραθυράκια έγινε μια ερώτηση. Τα παραθυράκια που αφήνουμε ανοιχτά. Κάθε κανόνας φυσικά πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά υπάρχουν πάντα παραθυράκια για να παρακάμψουμε τους κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε και να επιβάλλουμε τους κανόνες. Αυτό που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχων, ελέγχων σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν δηλαδή από τη μία ε, έλεγχη των ομοσπονδιών για να ελέγξουμε τι δουλειά κάνει κάθε επιμέρους ομοσπονδία ε, και πώς παρακολουθεί τις ποδοσφαιρικές ομάδες ομοσπονδία και επίσης υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί ε, επιθεώρησης, θα κάνουν audit, δηλαδή έλεγχο των ισολογισμών των ποδοσφαιρικών ομάδων και η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου με την Προεδρία του Jean-Luc έχει πάρα πολλές εξουσίες να ελέγξει, να επιθεωρήσει την οικονομική κατάσταση. Ε, είναι μια πρωτοφανής κατάσταση, πρωτόγνωρη και θα εφαρμοστεί από φέτος. Όλο αυτό το σύστημα των ελέγχων θα, προβλέψει, θα επιτρέψει, ελπίζουμε, σε μια αποτελεσματική λειτουργία και σε αποτελεσματικού ε, ελέγχους, ούτω ώστε να, να κλείσουν τα παραθυράκια. Αν συμβεί παρόλα αυτά αυτό, σε μια πρώτη φάση προβλέψαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ήπια, πειραματικού τύπου εργαλεία, να δούμε δηλαδή πώς πάνε τα πράγματα. Θα εντοπίσουμε ενδεχομένως ε, τις αδυναμίες, ή σημεία τα οποία αργότερα θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν θα μας επιτρέψει να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό. Ακούστηκε ένα σχόλιο για μια επόμενη πρωτοβουλία. για τα agency των ποδοσφαιριστών. Το σύστημα αδειών προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα ποσά που πληρώνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλους όσους βρίσκουν ποδοσφαιριστές. Υπάρχει υποχρέωση ε, οι ποδοσφαιρικές ομάδες να το κάνουν αυτό και αυτή η υποχρέωση θα αρχίσει να τρέχει από του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τα ξένα κεφάλαια, τι γίνεται με την εισαγωγή και την ροή ξένων, ξένων κεφαλαίων. Αυτό σίγουρα μας ανησυχεί, γιατί προφανώς βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι επωφελή, μπορεί να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Σίγουρα η ποδοσφαιρική ομάδα τονώνεται από την εισρωή αυτή ξένου κεφαλαίου, μπορεί να έχει άμεσες θετικές ε, αθλητικές επιπτώσεις, αλλά στο πιο ευρύ πλαίσιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ε, και μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα. Γιατί τι θα συμβεί, Φερρυπίν, αν από τη μία στιγμή στην άλλη οι ξένοι επενδυτέ αποσυρθούν, εξαφανιστούν. Υπάρχουν κίνδυνοι, όπω συνέβη και στο παρελθόν. Χρεοκοπία τη ποδοσφαιρικής ομάδα, με αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλες τι υπόλοιπε ε, ποδοσφαιρικές ομάδες. Δηλαδή, μιλάμε για μια καταστροφή σε ό,τι αφορά την ακαιρεότητα των διοργανώσεων. Τώρα, ένα σχόλιο που ακούστηκε για τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ποδοσφαιριστών θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, στοιχείο κλειδί. Εμείς προωθούμε όσο μπορούμε ε, και προτιμούμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες που ε, επενδύουν ε, στο να βγάλουν ένα ποδοσφαιριστή, στην κατάρτιση δηλαδή, παρά σε εκείνους που ψάχνουν να βρουν και να αγοράσουν. Επομένως, προσπαθούμε να πρημοδοτήσουμε τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων αυτών σε εθνικό επίπεδο, η UEFA εδώ δεν έχει αρμοδιότητε για την εφαρμογή των ιδίων αυτών κανόνων στα εθνικά πρωταθλήματα. Θεωρεί όμως ότι θα ήταν πολύ θετικό κάτι τέτοιο και ευχόμαστε οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες να εφαρμόσουν τις ίδιες αρχές αν όχι τους ίδιους κανόνες, τουλάχιστον τις ίδιε αρχές και για τη συμμετοχή σε εθνικά πρωταθλήματα. Υπ' αυτή την έννοια δουλεύουμε πολύ στενά με τις ενώσεις και τις ε, εθνικές ομοσπονδίες. Αυτό έγινε και για το σύστημα των αδειών. Όταν εισήχθη το 2004 το σύστημα των αδειών, οι ομοσπονδίες που το υιοθέτησαν σαν σε εθνικό επίπεδο ήταν πολύ λίγες. Ε, σήμερα είναι 45-53 και, τις ε, επόμενες δύο, και τα επόμενα δύο χρόνια θα φτάσουμε στα 49. 49 ομοσπονδίε 53. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αυτέ οι αρχέ τη καλή διαχείριση είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστούν έτσι με πολύ φυσικό και φυσιολογικό τρόπο και σε εθνικό επίπεδο. Un certain nombre de points διάφορα σημεία τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με το θέμα των αδειών ή το οικονομικό fair play. Για το anti-doping ε, είχε μια ερώτηση. Φυσικά εμείς εφαρμόσουμε τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά του ντόπινγκ. Ε, κάνουμε ελέγχους ε, μετά από κάθε αγώνα, αλλά και εκτός διοργανώσεων, με τρόπο έτσι ευνίδιο. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ευτυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένο σύστημα ντόπινγκ στο φούτμπολ. Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά κάτω του 0,1% στα τρία τελευταία χρόνια. Παραμένουμε άγρυπνοι όμως, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί όπως και στα άλλα αθλήματα και, το, και στο ποδόσφαιρο απειλούμαστε από αυτή τη μάστιγα. Και μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο για τα παράνομα στοιχήματα, τα οποία μας δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σήμερα. Και και αυτό το θέμα το έχουμε υπόψη μας. Ο Ιβο Μπέλετ μας μίλησε για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και της ισορροπίας των ε, διοργανώσεων. Τα βασικά έσοδα των ποδοσφαιρικών ομάδων προέρχονται από τα εθνικά πρωταθλήματά τους και όχι από τα, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι μύθος αυτό που λέγεται ότι τα χρήματα των ομάδων προέρχονται από τις ε, ευρωπαϊκές ε, διοργανώσεις. Προέρχονται κυρίως, κυρίως από τα εθνικά πρωταθλήματα. Όσο πιο ισχυρή είναι η, εθνική αγορά, τόσο πιο πλούσια είναι, πλούσιες είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες ε, συλλογικά ε, δίνουν τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Βέβαια, αλλάζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Υπάρχει μια μεγάλη ένωση στην Ευρώπη που έχει ένα σύστημα ατομικό για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και αυτή είναι η Ισπανία. Μας το υπενθύμισε ο Ισπανός συνάδελφο. Το να περιμένουμε ότι οι μεγάλε ισπανικές ποδοσφαιρικέ ομάδε θα αλλάξουν σύστημα ε, είναι, πολύ, είναι ουτοπικό. Είναι σαν να λέμε στις γαλοπούλες ε, να ευχηθούν να έρθουν γρήγορα τα Χριστούγεννα. Όχι, εξαρτάται από την Ομοσπονδία και από την Ισπανική Ένωση το τι θα γίνει. Δεν νομίζω θα κάνουν κάτι τέτοιο οι Ισπανικέ ποδοσφαιρικέ ομάδε. Τα επόμενα χρόνια ε, σκεφτήκαμε ότι έχει σημασία να δούμε πώ ε, μοιράζονται τα ωφέλη από τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, τα έσοδα από τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει που συνδέονται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και προφανώς εξαρτάται από τη σημασία της κάθε χώρας, δηλαδή ουσιαστικά τον πληθυσμό τη. Το ειδικό βάρος κάθε χώρας, άρα τον πληθυσμό της. Προφανώς, ε, οι ποδοσφαιρικέ ομάδες που προέρχονται από μικρές χώρες ε, μειονεκτούν σε σχέση με τις ποδοσφαιρικές ομάδες που προέρχονται από μεγάλες χώρες και όπου έχουν πολύ περισσότερου τηλεθεατέ, προφανώ αυτέ αυτές οι χώρες. Νομίζω ότι κάλυψε όλα τα θέματα περίπου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σουανί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι γνωρίζω κάπως τα πράγματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τόσο τέλεια αυτά τα πράγματα, όμως έχω δύο ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω αφενός όσον αφορά σε σχέση με τα όρια αυτά από την UEFA. Έχετε προβληματιστεί τι γίνεται σε σχέση με το αμερικανικό, ας το πω έτσι, πλαίσιο ανταγωνισμού και μετά το πλαίσιο της υπερχρέωσης. Ε, και ήδη στην αρχή είχε αναφερθεί αυτό το θέμα, ότι υπάρχει υπερβολική υπερχρέωση των ομάδων. Είναι υπερβολικά μεγάλος κίνδυνος αυτός. Και πάλι είναι κίνδυνος να χρησιμοποιήσει κανείς κάποια κόλπα γιατί δεν μπορεί να βγει από αυτή την κατάσταση υπερχρέωσης. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε στη συνέχεια και παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω και εγώ σε σχέση με την ΟΕΦΑ, θα προσπαθήσω ευχαριστώ για την παρουσίαση και εγώ θα ήθελα να πω ότι όπως ανακαλύφθηκαν τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν όπως και οι νότιες κυβερνήσεις των νότιων χωρών της Ευρώπης ανακάλυψαν δεν μπορούν να ζουν υπερχρεωμένες. Το ίδιο ισχύει και για τις ποδοσφαιρικές λέσχες. Σε σχέση με την ερώτηση της Προέδρου για τις ακυρώσεις ε, δεν δόθηκε μια ξεκάθαρη ε, απάντηση. Είπατε ότι ελπίζετε ότι θα μπορέσει να γίνει κάτι και ότι κάτι θα μπορούσε να επιτευχθεί με τις ε, κυρώσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σε βάθος, ιδιαίτερα όσον αφορά μεγάλες ομάδες και αισθάνονται ίσως ότι βρίσκονται ίσως εκτός αυτές θα ήθελα να θέσω εδώ δύο, να κάνω δύο παρατηρήσεις και σε σχέση με τους μισθούς ε, μία περικοπή, μία προσαρμογή είναι αναγκαία αν θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα και επίσης ε, να δούμε ότι κάποιες ε, ομάδες στην Ιταλία μπορούν να διαθέσουν τέτοιου είδους ποσά και όχι μόνο η περικοπή, η προσαρμογή των μισθών των ποδοσφαιριστών αλλά επίσης και των προπονητών Είχαμε ακούσει ότι για ένα συμβόλαιο υπάρχει ε, η δυνατότητα καταβολής 10 εκατομμυρίων ευρώ ετήσια και ίσως και κάνοντας λόγο για αυτά τα θέματα η χρονική ε, διάρκεια για τέτοιου είδους ε, μεταφορές για, από ένα, μία ομάδα στην άλλη θα πρέπει να μπορέσει να προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να δανειστεί εντός εισαγωγικών κάποιος παίκτη σε μια άλλη ομάδα και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, θα ήταν και δίκαιο κιόλας θα έλεγα και κατά τη διάρκεια της περίοδου και η πρόσληψη και απόλυση των προπονητών. Θα πρέπει αυτό σε σχέση με την, ε, τα όσα έχουν γίνει να εξεταστεί. Και ακριβώς αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση η οποία ε, δεν είναι πάρα πολύ καλή και δίνονται τέτοιες αμοιβέ μετά. Όλο το θέμα των συμβάσεων λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και να προσαρμοστούν τα πράγματα. Έχετε τα μέσα και την εξουσία για να επιβάλλετε αυτές τις προτάσεις. Ξέρω ότι θέλετε να το κάνετε και ξέρω ότι τα θέματα είναι δεδομένα και αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Αν όμως είναι να αντιμετωπιστούν, πρέπει να αντιμετωπιστούν, τότε σίγουρα οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι σαφέστατες και να είναι αποτρεπτικές και να είναι δεσμευτικές για να έχουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ε, Πολύ καλά κύριε Κέλλη. Θα σας στείλουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών για να έχετε κι εσείς αποτέλεσμα Κυρία Ντελά, Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι είναι επίκαιρη η έκθεση αυτή. Σε μένα ως Ολλανδία αφήνει μια επίγευση διότι ακούσαμε ότι από 38 επαγγελματικές ομάδες οι 14 ε, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι αυτό που παρουσιάσατε είναι ένα θεμητό μέσο για να ε, Επιτευθεί η εντυμότητα και η δικαιοσύνη ε, κατά τους αγώνες και, μεταξύ, και ανάμεσα σε αυτούς. Θα ήθελα να αναφερθώ στους, ε, στις παρεκκλήσεις. Αναφέρατε την νεότητα, την νεολαία, την, τα, τα κοινωνικά προγράμματα, αλλά ε, σκέφτομαι τις συνέπειες ε, εάν ε, αποτύχετε. Υπάρχει μια μικρή ομάδα στις κάτω χώρες, δεν είναι πασίγνωστη ομάδα, είναι κοντά στην περιοχή που μένει η αδερφή μου, αλλά η ομάδα αυτή συνάντησε πολύ μεγάλες δυσκολίες επειδή επένδυσε σε μεγάλο στάδιο σε τελείως ακατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα της υποδομής και μια γενική ερώτηση προς τον κύριο Γκαγιά που είπε ότι όσο πιο μεγάλοι οι αγώνες, τόσο πιο πλούσιες οι ομάδες, άρα, άρα θεωρητικά και ε, περισσότερη οικονομική ευρωστία. οι κάτω χώρες ε, εργάζονται σκληρά διότι ε, θα ε, δεχτούν τους παγκόσμιους αγώνες το 2018. Αλλά εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Πολλές παρατηρήσεις ακούτε. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε σήμερα ήταν κάποιος πιο θεωρητικά, αλλά μπορεί η UEFA να έχει εκπονήσει πολύ πιο συγκεκριμένο σχέδιο, πτώση όσον αφορά ε, ε, το, το, ε, την αρνητική οικονομική κατάσταση Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να υποχρεώσουμε τις ομάδες ε, να μην έχουν ε, σημαντικά ελλείμματα. Τίθεται το θέμα τότε του ισοσκελισμού των λογαριασμών τους. Τι γίνεται με τους παίκτες όταν μεταγράφονται Υπάρχουν ε, οι λογαριασμοί εκπονούνται σύμφωνα με τους ίδιους ε, κανόνες και ελέγχονται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Αλλιώς δεν έχει ε, νόημα να θεωρήσουμε το έλλειμμα απλά ένα από τα απαραίτητα κριτήρια. Εάν ε, λοιπόν ε, ε, ισοσκελίζονται με τον ίδιο τρόπο οι λογαριασμοί, εάν ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο οι λογαριασμοί, αυτό θα με ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δω τι συνέπειες θα έχει. διότι αλλιώς μπορεί να βλέπουμε όλο και περισσότερο δανεισμό των ομάδων ε, και ε, τα ελλείμματα προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παίκτες ε, πληρώνονται περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει η ομάδα. Λοιπόν, μήπω θα έπρεπε να σκεφτούμε και το θέμα αυτό πρώτου περιορίσουμε τις αμοιβέ των παικτών. Άλλωστε υπάρχουν χορηγοί που αναλαμβάνουν μέρος του, κόστους του κόστους. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αναγκάζουμε, θα αναγκάσουμε τις ομάδες να εφαρμόσουν ε, τα μέτρα αυτά. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν ε, ε, μία νυχτή, αλλά ποιος είναι ο στόχος. Διότι ένας από τους στόχους μας είναι η ανταγωνιστικότητα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρότσμαν και κυρία Um, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα να μας παρουσιάσετε τις θέσεις σας. Έχω κάποιες ε, ανησυχίες σχετικά με το αν έχετε πετύχει την ε, σωστή ισορροπία. Θα ήθελα λοιπόν, λοιπόν να σας ρωτήσω ε, κάποια πράγματα. Αποκλείονται πολλές μεγάλες ομάδες με τα μέτρα σας ε, αυτό δεν θα ε, είναι εις βάρος της ποιότητας των ε, αγώνων. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πολλές μεγάλες ομάδες. Ακούστηκαν από άλλα μέρη της Ευρώπης επιφυλάξεις κατά διάρκεια των διαβουλεύσεων που είχατε και επίσης μπορείτε να αναφερθείτε στα best ownership models, στα ε, μοντέλα ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ. Κυρία Μακλάκη, νομίζω ότι δεν κατάλαβα σωστά. Είπατε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη. Ε, το και μάλλον δεν είναι σωστό. Η κυρία Χάνιμπαλ. θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ σε αυτό. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το ποδόσφαιρο. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα ίδια πράγματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε το σήμερα να κάνετε την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θέλω να φανώ αρνητική ή απεσιόδοξη, αλλά αυτά που είπατε ακούγονται πολύ ωραία για την πλειοψηφία των ομάδων, αλλά θα ήθελα πολύ να μου πείτε τι ισχύει για τις ομάδες σαν την Chelsea ή την Manchester United. Ε, πώς θα εισαχθούν στο σύστημα αυτό. Και γενικά ποιος είναι ο στόχος μας. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας, διότι φαίνεται ε, ότι για τις ε, πλούσιες αυτές ομάδες, που δεν είναι όλες βρετανικές, ότι εφαρμοστεί σε αυτές φαίνεται ότι θα έχει συνέπειες και για τις άλλες ομάδες. Θα υπάρχει η φιλοδοξία να φτάσουν οι ομάδες στην κορυφή και μπορεί συχνά να ξεπεράσουν τις δυνατότητές τους ε, για να το πετύχουν αυτό. Προσπαθούν να φτάσουν στα ανώτερα επίπεδα και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Αυτό δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό. Έχετε λοιπόν να παίξετε σημαντικό ρόλο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Μιλάμε για συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, για ε, ανταγωνιστική ισορροπία. Είναι πολύ δύσκολο όμως να εξετάσουμε ρεαλιστικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Λίγο πιο θετική να είμαι να ρωτήσω τι έχετε να πείτε για την ε, προπόνηση των ε, παικτών. Ε, μιλήσαμε για την προώθηση νέων παικτών από τις ομάδες. Το σύστημα όμως και πάλι είναι μάλλον αποθαρρυντικό, διότι εφόσον μπορεί να αγοράσει κανείς αλλοδαπούς παίκτες, αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα επενδύουν λιγότερο στην δική τους προπόνηση, στην προπόνηση των νέων νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί, το, ο τρόπος που προτείνεται μπορεί να παρακάμψει το πρόβλημα, αλλά όχι να το λύσει απόλυτα. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. the discussion is ended and I... Έληξε η συζήτηση. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Γκαγιά ή τον κύριο Τραβέρσο να απαντήσουν. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω από τα μη οικονομικά θέματα και ο συνάδελφός μου θα σας διαφωτίσει για τα αμυγός οικονομικά θέματα. Το θέμα των ε, ποδοσφαιρικών ομάδων που είναι πολυεθνικές, ας πούμε τις Μπενελούξ. Δεν τίθεται μόνο για τον Μπενελούξ, αλλά για την ε, Κεντρική Ευρώπη, για την πρώτη Ιουγκοσλαβία, για την πρώην ε, Σοβιετική Ένωση, για τη Σκανδιναβία υπάρχουν τέτοιες ομάδες πολυεθνικές ας πούμε, περιφερειακές. Κάντε μα προτάσει είναι η θέση μα. Εάν ε, συμφωνούν οι ομοσπονδίε ε, και οι ποδοσφαιρικέ ενώσει, μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μα. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε ε, προσαρμογές για το πώς θα έχουν πρόσβαση στι Ευρωπαϊκέ διοργανώσει αυτέ οι ποδοσφαιρικέ ομάδε αλλά αυτέ οι ομάδε με τι ομοσπονδίε του θα πρέπει ατομικά να έρθουν να μα πούν, να πούνε θέλουμε να συγχωνευτούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ποδοσφαιρική πολυεθνική ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ό,τι αφορά του ποδοσφαιριστέ που καταρτίζονται ε, στη χώρα του, τοπικά α πούμε, από τη στιγμή που έχουμε εισαγάγει το μέτρο, διάφορες εθνικές ομάδες ε, το υιοθέτησαν ε, μια και είσαστε Αγγλίδα, πρέπει να σας πω ότι στην Αγγλία υπάρχει αυτό το μέτρο για την ε, τοπικών παιχτών και το οικονομικό fair play δεν έχει άμεση σχέση με αυτό το ζήτημα. Αλλά το οικονομικό fair play ε, δίνει τις δυνατότητες να... και, και κάποια πλεονεκτήματα για να επενδύσουμε στην κατάρτιση των νέων στην προπόνησή τους και στην κατάρτισή τους παρά στην αγορά τους. Και αν το συνδυάσουμε με τους κανόνες προνομίων για παίχτες που έχουν καταρτιστεί και προπονηθεί ας πούμε, τοπικά, α, όντως δίνουμε, χωρίς να επιτάσουμε, χωρίς να επιβάλλουμε, ας πούμε, κάποιες, κάποια κίνητρα στις ποδοσφαιρικές ομάδες για να το κάνουμε Ακούστηκαν μια σειρά από σχόλια και ερωτήσεις για το ανώτατο όριο των αποδοχών των αμοιβών των ποδοσφαιριστών κατά το αμερικανικό μοντέλο. Εμείς πήγαμε στις ΗΠΑ πάνω από ένα χρόνο πριν ε, με τον Τζάνι Φαντίνο, ε, το Γενικό Γραμματέα, ε, για να δούμε τα διάφορα μοντέλα ανώτατου ορίου των αμοιβών. Γιατί δεν είναι όλα τα ίδια που εφαρμόζονται στις διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες των ΗΠΑ. Και συνειδητοποίησαμε πάρα αυτό το αμερικανικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό από το ευρωπαϊκό. Έχει και μια μεταφορά αυτού του ανώτατου ορίου των αποδοχών ε, από την Αμερική στην Ευρώπη θα ήταν πολύ περίπλοκο ζήτημα. Όταν μιλάμε για την UEFA, μιλάμε για 53 ομοσπονδίες που είναι μέλη της UEFA. Μερικές από αυτές, περίπου οι μισές, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιπε περίπου το 50% δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, να φτάσουμε στους ίδιους στόχους, μέσα όμως από μονοπάτια και οδούς λιγότερο επιτακτικούς, λιγότερο παρεμβατικούς. να μην παρεμβαίνουμε στο πώς ε, γίνεται η διαχείριση ε, της ομάδας. Να μην πούμε θα πρέπει να μειώσετε τόσο τους μισθούς, ας πούμε, τόσο τα 100. Λέμε, θα πρέπει να λειτουργείτε με τα έσοδά σας. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάποια δαπάνες αναγκαστικά θα πρέπει να μειωθούν. Και επειδή οι πιο σημαντικές δαπάνες είναι οι μισθοί και οι μεταγραφές, αμα, αυτόματα οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν ένα σοσκελισμό με βάση αυτά τα, αυτές τις δύο βασικές δαπάνες. Μισθή δηλαδή και μεταγραφές. Φυσικά θα υπάρχουν ε, και στο μέλλον ε, ποδοσφαιριστές στάρ που θα πληρώνονται εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα, πληρώνονται, θα καταβάλλονται εκατομμύρια για τη μεταγραφή τους. Το βασικό όμω είναι να μπορούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες να τιμήσουν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά τα χρέη, 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου είναι το συνολικό χρέος. Ε, σημαντικό ποσό. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να αυξηθεί έτσι περαιτέρω αυτό το χρέος. Γιατί στα πλαίσια του ισοσκελισμού, του ισολογισμού, τα... οι τόκοι που πληρώνονται για το χρέος λαμβάνονται υπόψη. Και αν ένα... και μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν μπορεί να πληρώσει το χρέο της, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διοργανώσει μας. Γιατί δεν λειτουργεί με τρόπο δίκαιο. Δεν σέβεται το fair play. Δεν παίζει δίκαια, αν θέλετε. Επίσης, έγινε λόγος για τις εξαιρέσεις, για τις υποδομές, επενδύσεις στις υποδομές. Αν επενδύσει κάποιος σε αθλητική εγκατάσταση, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτή είναι μια τεράστια επένδυση και μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες οικονομικές για την ομάδα. Όπως είπα, αν γίνει, γίνουν επενδύσει σε ένα στάδιο ε, και υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα, τότε συσσωρεύονται ε, τόκοι που θα πρέπει να πληρωθούν και πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ισολογισμού της ομάδος. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις που, που αφορούν τα μη οικονομικά, α, τις μη οικονομικές δαπάνες, δηλαδή η απόσβεση των, ε, υποδομών που, πρέπει, που μπορούν να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό. Αλλά είναι κόστος μη οικονομικό, μη νομισματικό αν θέλετε. Ο κύριος Κρόιτσμαν αναφέρθηκε σε κανόνες reporting, αναφορών, που δεν είναι ίδιες όλες τις χώρες. Πρέπει όμως να είναι ίδιες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι προσφυγικές ομάδες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, λειτουργούν με την ίδια μεθοδολογία. Οι κανόνες μας προβλέπουν ε, κανόνες για τις αναφορές οι ίδιους και ελέγχους που γίνονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα. Πέρα από το ότι δημιουργήσαμε αυτή την Επιτροπή Ελέγχου που ήταν εξάρτητη σε υπερεθνικό επίπεδο, γιατί αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που βασίζονται στην ε, διοίκηση και στο οργανόγραμμα της ΣΟΕΦΑ και θα κάνουν μια σειρά από ελέγχους. Αυτό θα μας επιτρέψει, αυτή η Επιτροπή δηλαδή, θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα επίπεδο ελέγχου και αποπτίας εντελώς ανεξάρτητης και θα εξασφαλίσουμε μία ενιαία εφαρμογή των κανόνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Την ίση μεταχείριση, το equal treatment όλων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ακούστε κανένα σχόλια και ερωτήσεις για την κατάσταση κυρίως στην Αγγλία. Ένα ερώτημα ακούστηκε για το καλύτερο δυνατό μοντέλο επιχειρηματικό, εταιρικό για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο ιδανικό, ιδα, ιδεατό. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα. Σε στατιστικό επίπεδο είδαμε ότι στην Ευρώπη περίπου το 50% των ποδοσφαιρικών εταιριών δεν είναι η κατάλληλη λέξη αυτή, καλύτερα να τις, ομα... να τις ονομάζουμε ποδοσφαιρικές ομάδες, είναι associations, είναι οργανώσεις. Οι υπόλοιπε είναι εταιρείε. Είναι μετοχικές εταιρείε, ανώνυμες εταιρείε. και δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση της ομάδας αυτή, που, της αθλητικής ομάδας δηλαδή, όπου συμμετέχει στις αγώνες, στις διοργανώσεις κτλ. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτέ οι εταιρείε. Οι ποδοσφαιρικέ ομάδες, ανεξάρτητα από τη δομή τους, θα πρέπει να την χάνουν ε, δημοκρατικής και διαφανούς διαχείρισης. Το σύστημα των αδειών θέτει ένα σύστημα, ένα, μια δέσμη από κριτηρίων, μια δέσμη κριτηρίων ακριβώς για, για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Εμεί θεωρούμε ότι χάρη σε αυτού τους κανόνες θα υπάρχουν διοργανώσεις πιο ποιοτικέ. Θα εφεληθούν οι διοργανώσεις από τους κανόνες ελέγχου ε, πιο επιτακτικού. Δεν θα πληγούν αντίθετα οι διοργανώσεις. Ε, θα εξασφαλιστεί μία βιωσιμότητα. Ελάχιστες είναι είναι διά, διάφορες συγγνώμη, οι ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες ε, κήρυξαν πτώχευση κατά τη διάρκεια α, μίας διοργάνωσης. Ε, όλη η διοργάνωση ε, επλήγει από αυτό το γεγονός. Επομένως είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Πολύ σημαντικοί αυτοί οι κανόνες. Σήμερα οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην Ευρώπη. Αν ένας παίχτης ε, παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και αύριο μεθαύριο ε, παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ maximum, δεν νομίζω ότι θα πληγεί η ποιότητά του. Ο παίχτη είναι παίχτη και παίζει με τι ικανότητέ του. Δεν νομίζω ότι θα έχει επιπτώσει λοιπόν η μείωση του μισθού του στην ποιότητα του παιχνιδιού του. Η κατάσταση που βρισκόμαστε είναι πια. Είναι η εξή. Υπενθυμήθηκε, υπενθυμίστηκε προηγουμένω ότι πολλέ ε, ομάδες, ε, όχι της πρώτης εθνικής, κατώτερων ε, εθνικών, μικρομεσαίες, στην προσπάθεια να πλησιάσουν τις μεγάλες σούπερ ποδοσφαιρικές ε, δυνάμεις, παίζουν, συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά στοιχήματα. Αυτή η κερδοσκοπική και παράλογη στάση ε, ενέχει κινδύνους. Και όταν δεν υπάρχει επιτυχία, ε, και ξέρετε, στο ποδόσφαιρο ένας κερδίζει, όχι και δύο ομάδες, τότε η κίνδυνη για την εν λόγω ομάδα είναι τεράστια. Έχουμε έσοδα τότε που παίζουν ανάλογα με τα αποδοσφαιρικά αποτελέσματα, αλλά το κόστος δεν παίζει καθόλου για αυτή την ομάδα, γιατί είναι δεδομένο για μια χρονική περίοδο 3 με πέντε χρόνια. Δηλαδή παίζουν, στοιχηματίζουν συστηματικά για τη συγκεκριμένη περίοδο, το κόστος είναι δεδομένο, το αποτέλεσμα όμως αλλάζει. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν ε, μπορεί να προβλέψει πάντα τον νικητή. Εμείς θέλουμε, λοιπόν, να, μέσω του συστήματος που σας περιέγραψα, να προωθήσουμε μια συμπεριφορά πιο ορθολογική. Η, τα στοιχήματα για το ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα θα περιοριστούν και θα υπάρξει μια μεγαλύτερη σταθερότητα. Θεωρούμε ότι το χάσμα ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μειωθεί. Γιατί τα τεράστια ποσά που δίνουν οι μεγάλοι μέτοχοι στο μέλλον αναγκαστικά θα μειωθούν ή θα πάρουν άλλη κατεύθυνση. Θα πάνε σε, βραχυ... σε μακροπρόθεσμες ε, και μακροχρόνιες επενδύσεις. Επομένως το χάσμα θα μειωθεί. Ας ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τους κυρίους Τραβέσο και Γαλιά για το ότι ήταν εδώ παρόντες ε, και για τα όσα μας εξέθεσαν με τις εισηγήσεις τους και ελπίζουμε φυσικά ότι αυτά τα οποία συλλάβατε και προτείνατε θα είναι σε κάποιο βαθμό εφαρμόσιμα. Χρειάζεστε ανθρώπους που θα ακολουθήσουν τις προτάσεις σας και θα προσαρμοστούν σε αυτές. Και χρειάζεστε και για την εποπτεία ένα μηχανισμό, έναν ανεξάρτητο μηχανισμό. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Και αν σκεφτώ τον κύριο Κρότσμαν και την κυρία Ντελάνια για τα όσα ανέφεραν και έθιξαν, το θέμα ποια στοιχεία θα, έχουν, θα υπάρχουν ως βάση και πώς θα εξετάζονται τα οικονομικά, με ποιο τρόπο όλα αυτά θα ελέγχονται τελικά. Ε, τότε έχουμε ένα μεγάλο πλέγμα, ένα πολύ μεγάλη δουλειά μπροστά σας. Εσείς έχετε αυτή τη δουλειά, πρέπει να την επιτελέσετε. Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι όλοι με ιδιαίτερη προσοχή θα παρακολουθήσουν αυτά τα τεκτενόμενα και προς το συμφέρον σας και των παικτών και των μικρότερων λεσχών. Ελπίζουμε ότι αυτά θα γίνουν πραγματικότητα, όχι τον επόμενο χρόνο, αλλά στα επόμενα δέκα χρόνια. Και πάλι σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε θερμά. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάρκεια. Και περνάμε έτσι στη συνέχεια στο σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Πού είναι ο κύριος Μπέλετ. Λοιπόν, έρθει να καθίσει. Περνάμε λοιπόν, λέω... Ζητώ από όλους παρακαλώ να περάσουμε στο επόμενο σημείο αν θέλετε. Okay. Εντάξει, περνάμε στο σημείο εξή στην ημερήσια διάταξη. Κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα για την ψηφιακή εποχή, το μέλλον ε, του διτού συστήματος, dual system. Ιβο Μπέλετ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thanks very much. Θα ε, ε- σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα δώσω μια σύντομη εισαγωγή. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων και θα αφήσω όσο το γίνεται μεγαλύτερο περιθώριο για να συζητηθούν τα πράγματα, να γίνει μια συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είχαμε πολλές επαφές στις τελευταίες πρόσφατες εβδομάδες με πολλούς εμπλεκόμενους ε, και μετέχοντες ε, και ο κατάλογος των επαφών είναι στα έγγραφα, σχεδόν όλοι αναφέρονται εκεί. Δεύτερον, να αναφέρω επίσης το γεγονός ότι ήδη είχαμε μία πρώτη καρποφόρα επαφή με ε, τους περισσότερους κοιόδης εισηγητέ των κοινοβουλευτικών ομάδων, πράγμα που είναι σημαντικό για να έχουμε το δυνατόν περισσότερες προτάσεις ως input από όλες τις πολιτικές ομάδες που είναι παρούσες εδώ, να υπάρχει μια μεγάλη πλατφόρμα και υποστήριξη για αυτή την έκθεση και ελπίζω φυσικά ότι θα σημειωθεί πρόοδος με τον ίδιο επικοδομητικό τρόπο. Λοιπόν, απλά δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω, κυρία Πακ. Πρώτον, να υπενθυμίσω και πάλι ποιο είναι το εύρος, ο στόχος αυτή της έκθεση. Τι εντάσσεται στον τίτλο είναι σαφές, αλλά είναι φυσικά και σημαντικό να το τονίσουμε, ότι εδώ πρόκειται για το μέλλον του διπλού, διτού συστήματος. Διτού υπάρχουν δύο εταίροι δηλαδή. Το δημόσιο κρατικό τομέα, τομέας αφενός και ο εμπορικός των ιδιωτών αφετέρου. Και αυτό είναι κάτι το μοναδικό για την Ευρώπη. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις είπα. Με αυτό το διτό σύστημα το οποίο έχουμε πολύ κοντά στην, μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε να έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του κρατικού τομέα στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και του ιδιωτικού τομέα, εμπορικού τομέα φετέρου. Να υπενθυμίσω λοιπόν εδώ κάτι σε σχέση με τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που έχουν ε, εγκριθεί από τους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης που θα έλεγα ότι είναι σημαντικά θέματα και μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε ως βάθρα για να χτίσουμε σε αυτή τη βάση. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την διοργάνωση των ε, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ε, τα τελευταία χρόνια και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν την ανεξαρτησία των κρατικών τηλεοπτικών σταθμών, σημαντικό στοιχείο αυτό και αυτό συνδέεται πολύ κοντά με την χρηματοδότηση και την εγγυημένη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αυτών των τηλεοπτικών εκπομπών που πρέπει να διευκολύνεται και μέσω ενός διαρκού σχεδιασμού και προγραμματισμού όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που προτάθηκαν από το Συμβουλίο της Ευρώπης. Και πάλι τώρα εδώ δεν είναι στόχος μας, δεν είναι πρόθεση αυτής της έκθεσης του εισηγητή αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή, να προσπαθήσουμε να αναμειχθούμε και να ε, παρεύουμε σε εθνικέ αρμοδιότητε. Γνωρίζουμε πολύ καλά το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ που πάλι τονίζει την αρχή τη επικουρικότητα και το γεγονό ότι κατά μεγάλο βαθμό αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι εθνική αρμοδιότητα. Και δεν θέλουμε να αναμειχθούμε ή να αμφισβητήσουμε, να υπονομεύσουμε αυτή την σημαντική αρχή. Όμως από την άλλη πλευρά θα έλεγα, πιστεύω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το ότι πρέπει απλά να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις ε, υπέρ αντιστάθμισης όπως έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν και εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να εξετάσουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει απουσία χρηματοδότησης, έλλειψη χρηματοδότησης και όπου υπάρχει το θέμα της ε, ε ανεξαρτησίας των εκπομπών. Είναι δουλειά μας να τονίσουμε τα, προβλήματα που ίσως υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν σίγουρα έχουμε απέναντί μας και αυτό αναφέρεται και στο εύρος και στον τίτλο της έκθεσης έχουμε απέναντί μας έναν με πολύ κατακαιρματισμένο τομέα ε, εκπομπών και ε, μεντιακών μέσων, μέσων ΜΜΕ και έχουμε εδώ μεγάλους εμπλεκόμενους και παίκτες παράλληλα με τους παραδοσιακούς σταθμούς ε, Telecom, ε, έχουμε τους παρόχους, ε, έχουμε citizen journalism, να χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες αυτού του είδους δημοσιογραφίας που αναπτύσσεται και βρίσκεται υπό, εξέλιξη καθημερινά και που είναι πρόκληση για τα παραδοσιακά μέσα <clears throat> ακόμα και για τον έντυπο τύπο, τον γραπτό τύπο φυσικά. Μέσα σε αυτό το νέο περίγυρο πλαίσιο και περιβάλλον οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να δούμε ότι σχεδόν μειώνονται, φθήνουν και φιλορωούν και σχεδόν εξαφανίζονται. Και αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα και νομίζω μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Αυτό οδηγεί σε έναν όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο τέλος τέλος μεταξύ των κρατικών δημόσιων μέσων αφενός και του διαδικτύου και των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και από την άλλη πλευρά των ε, εκδοτών, περιοδικών και εφημερίδων και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, και αυτό είναι μία από τις κυριότερες προκλήσεις, όχι μόνο σε αυτήν την έκθεση, αλλά και σε όλο το εθνικό επίπεδο και σε όλους τους εμπλεκόμενους στα ΜΜΕ, στα κράτη-μέλη και τους ε, υπεύθυνου για την πολιτική. Θέλουμε να υπάρχει ένα ισόρροπο με, μέτρο συμβίωσης και των δημόσιων αλλά και των, των δημόσιων και των ιδιωτών και των εκδοτών του γραπτού τύπου και των περιοδικών και εφημερίδων και όσων ε, μετέχουν σε τέτοιου είδους ε, εκπομπές ε, τηλεοπτικά και όλους όσοι συμμετέχουν και στο διαδίκτυο για να υπάρχουν αϊφότυπα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να υπησέθω σε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρυσι όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις και την εφαρμογή αυτού του πλαισίου σημαντική υπόθεση σε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι όταν οι δημόσιοι, δημόσιες ε, ε, τέτοιες εταιρείες θέλουν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες ε, ψηφιακά, ότι αυτό θα πρέπει να συνάδει και να ταυτοποιείται και να υπάρχει μια αξιολόγηση αυτών των πρωτοβουλειών. Τα γνωρίζουμε αυτά από πέρσι ήδη. Και πάλι δεν είναι η πρόθεσή μας εδώ, δεν είναι η πρόθεση του εισηγητή και ούτε και η πρόθεση θα έλεγα και αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να ανανεώσουμε ή να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση όσον αφορά την ανακοίνωση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν είναι αυτός ο στόχος αυτής της ε, έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Και στρεφόμενος τώρα σε κάποιες από τις προτάσεις. Προτάσεις ε, για το μέλλον. Επιτρέψτε μου πρώτα να πω ότι, η μία κοινή προσέγγιση για όλους, one size fits all, δεν είναι κάτι το εφικτό, γιατί είναι ισοπεδωτική προσέγγιση. Η κατάσταση στη Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο Βέλγιο είναι τελείως διαφορετική από την κατάσταση στη Σλοβακία, Ρουμανία ή Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να έχουμε λοιπόν εξειδικευμένε χειροπιαστέ λύσει για ιδιότυπε καταστάσει με τι ιδιομορφίε του. Για να είμαι πιο χειροπιαστό και συγκεκριμένο, δεν θα απαριθμίσω όλα όσα έχουμε προετοιμάσει εδώ. Έχει διανεμηθεί ήδη ένα σχέδιο πρόταση πρότασης ψηφίσματος σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εδώ παρόντα και ηλεκτρονικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και ε, γραπτός. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ή τρία συγκεκριμένα πιο εξειδικευμένα στοιχεία του σχεδίου ψηφίσματος που προετοιμάσαμε και θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας φυσικά στις επόμενες εβδομάδες. Πρώτα απ' όλα και κύρια το σημείο 8 και το σημείο 9. Τι λένε αυτά. Λοιπόν, αυτά λένε και υπενθυμίζουμε σε αυτά τα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω είναι σημαντικό, υπενθυμίζουμε σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις δεσμεύσεις που έχουν ε, αναλάβει όσον αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα των ε, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Αναφέρομαι στις συστάσεις και κατευθυντήριες ε, γραμμές που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς ως Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχέση με την επικουρικότητα, πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να σέβονται αυτές τις δεσμεύσεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή επιτόπου καθημερινά και ζητάμε, και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο, και αυτό είναι ένα στοιχείο που ε, λέει το εξή. Ζητούμε με τη δική σα σύμφωνη γνώμη φυσικά. Είναι σχέδιο ψηφίσματο, σχέδιο πρόταση. Στοχεύουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να δώσουν σαφείς ε, ε, ε, εντολέ με συγχωρείτε στο παρατηρητήριο του Στρασβούργου, Στρασβούργου να επιτηρεί τον τρόπο, να εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σε αυτές τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνήσει ήδη μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και των προτάσεών του. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία αυτής της πρότασης ψηφίσματος που είναι σημαντικό. Ένα άλλο Προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες τώρα από όσα έχουμε συντάξει. Δεν προσπαθώ να αναγνώσω όλα όσα έχουμε ενώπιόν μας. Ένα άλλο θέμα από το έγγραφο και που θέτουμε υποσυζήτηση απόψε είναι Θέλουμε να ζητήσουμε και να ενθαρρύνουμε από όλους τους εμπλεκόμενους και μετέχοντες μέσα στις ε, επαφές μας για την ψηφιακή αυτή δράση να συνεργαστούν από κοινού στενά. Έχουμε διάφορα παραδείγματα ήδη, συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων τέτοιων ε, συνεργασιών που υφίστανται. Αναφέρομαι ήδη στο BBC όπου υπάρχουν πολλές ανταλλαγές ε, όσον αφορά οπτικοακουστικό υλικό μεταξύ BBC αφενός και εκπροσώπων <clears throat> του γραπτού τύπου εφημερίδων ε, και περιοδικών, τέτοιου είδους ανταλλαγές οπτικοακουστικού υλικού. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια σωστή πορεία, καλή οδός να πορευτούμε προς το μέλλον, να οδεύσουμε προς το μέλλον και ζητούμε, στοχεύουμε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία. Όχι νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά να δώσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να συνέλθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στα μίντια, στα ΜΜΕ, για να υπάρξει μια αηφορία όσον αφορά τα πρότυπα των ανταλλαγών αυτών οπτικού ακουστικού υλικού μεταξύ των ε, ε, μέσων και να λάβουμε υπόψη τα πρότυπα που υφίστανται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο αυτά, αλλά και πρότυπα που υφίστανται βέλτιστων πρακτικών και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Λοιπόν, εν κατακλείδη συνοψίζοντας, υποσχέθηκα θα είμαι σύντομος Πρόεδρε. Νομίζω είναι κέρια σημασία. Κύριο θέμα να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον και ως κοινωνία έχουμε την προοπτική νομίζω και ως κοινοβούλιο να βοηθήσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να αποφύγουμε το ψηφιακό έλλειμμα το ψηφιακό χάσμα, ας το αποκαλέσω έτσι, μεταξύ εκείνων που θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο αφενός και εκείνων των πολιτών αφετέρου που δεν θα έχουν πρόσβαση ή προσπελασιμότητα σε αυτά τα στοιχεία, δεν θα έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία αυτά στο διαδίκτυο. Θα έχουμε δηλαδή τους έχοντες και κατέχοντες ψηφιακά και τους απόρους μη έχοντες από την άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει να υπάρχει μέγιστη προσπελασιμότητα και εύκολη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Και για να ολοκληρώσω και για να αναφερθώ και στην πρόεδρο ακριβώς αυτής της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής παράθεμα. Δεν ήταν στατικό προϊόν το ψηφιακό αυτό εγχείρημα, αλλά μία ενεξελίξη διαδικασία. Εν μια διαδικασία σε διαρκή πρόοδο και μετεξέλιξη. Πάντα ρί λοιπόν. Αυτά ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Κύριε Κέρκχοπ θα ξεκινήσετε και θα συνεχίσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Απογοητεύομαι λίγο που έπρεπε να φύγει η πρόεδρος της Επιτροπής μας, διότι Ελπίζα να ακούσω την απάντησή της. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε ε, στη Βρετανία και το υπόλοιπο της Ευρώπης. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να ε, δείτε το διαγωνισμό της Eurovision που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Ε, ο διαγωνισμός αυτός έδειξε για άλλη μια φορά ότι η Βρετανία απήχε από το υπόλοιπο της Ευρώπης. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο για το εξαιρετικό έγγραφο εργασία. Δεν θέλω να τονίσω πολύ την ηλικία μου, αλλά προέρχομαι... Η εποχή μου ήταν η εποχή που έπρεπε ε, το, η, ιδιωτική ραδιοτηλεόραση να ε, αγωνιστεί για να πετύχει τη θέση, τη θέση της. Ε, είμαι ε, πρόεδρος ε, ενός δικτύου ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο, στη βορειοανατολική Αγγλία. κάποτε είμαστε, λειτουργούσαμε πειρατικά, δίναμε στους νέους αυτό που δεν μπορούσαν να βρούνε από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που ήταν βαρετά και σαν φάρμακο που δεν έχει καν ωραία γεύση. Και αυτό θα ήταν άλλωστε το φάρμακο τώρα. Θα δεχόμασταν ε, ότι κάποιοι ε, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί είναι απαραίτητοι, αρκεί να, το φάρμακο να έχει ευχάριστη γεύση. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο συνάδελφος ε, είναι σωστό όσον αφορά την ενιαία προσέγγιση για όλους. αυτό δεν είναι ε, εφικτό, διότι ε, σε κάποια κράτη-μέλη η ιδιωτική ε, ραδιοτηλεόραση είναι πολύ ανεπτυγμένη, σε άλλες όχι. Οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται, βλέπουμε αυξανόμενο ανταγωνισμό και η διαφήμιση είναι η απαραίτητη διαδικασία χρηματοδότησης. Είδαμε επίσης κρατική, την κρατική ραδιοτηλεόραση να μπαίνει σε τομείς όπου δεν πληρεί τα κριτήρια. Δηλαδή τομείς που μπορούν ε, κάλλιστα να εξυπηρετηθούν από ε, ε, την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, χρειάζονται όμως, θεωρούν ότι χρειάζεται να ανταγωνιστούν στον τομέα αυτό, διότι θέλουν να έχουν τον έλεγχο για ε, το τι εκπέμπεται. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ ε, σχετικά με το πώς θα επιτρέψουμε να εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στη, στους ιδιωτικούς και στους δημόσιους ε, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ όσον αφορά τους ορισμούς. Επιτρέψτε μου να να πω όσον αφορά την εισαγωγή στην αγορά. Κάποια ιδιωτικά κανάλια θεωρούν ότι το σύστημα που υπάρχει ε, τους έχει ε, εμποδίσει να εισέλθουν. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα λοιπόν για να περιορίσουμε την ε, ένταξή τους στον χώρο αυτόν. Μια υπηρεσία αδειοδότησης θα πρέπει να ενεργεί για το κοινό όφελος. Όσον αφορά την ψηφιακή ραδιοφωνία και τα μη ψηφιακά προγράμματα. Έχω μια ηλικία, μπορεί να μην θυμάμαι την κατάσταση ε, στην Ουγγαρία το 1956, θυμάμαι όμως ε, την άνοιξη της Πράγας το 1967, όταν το ραδιόφωνο ήταν ο μόνος τρόπος ε, να μάθει ο κόσμος για τα φρικτά πράγματα που εκτιλήσονταν τότε. Τώρα όμως ε, βλέπουμε ότι πολλά κανάλια εμποδίζουν τον κόσμο να ε, βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο. Δεν θέλουμε λοιπόν τα τεχνικά μέσα να παρεμποδίσουν ε, την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω όλο και περισσότερο την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και θα ήθελα να τονίσω ότι Όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών αυτών από το διαδίκτυο, ναι, υπάρχει εδώ προτεραιότητα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φροντίσουμε το διαδίκτυο να μην ε, παρέχεται μόνο σε κάποιους προνομιούχους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές. Για να έχουμε ελεύθερη ευρυζωνική πρόσβαση, θα πρέπει να φροντίσουμε όλες οι ε, κυβερνήσεις ε, στην Ευρώπη να στηρίξουν τα μέτρα αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα μαζικό πρόγραμμα για να παρασχεθεί ευρυζωνική πρόσβαση σε υπαίθριες περιοχές που στο παρελθόν δεν είχαν τέτοια πρόσβαση. Ελπίζω λοιπόν έτσι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ακολουθεί στην κατεύθυνση αυτή. Θα υποβάλει προτάσεις ε, Ξέρω ότι τώρα απλά κάνουμε μια αρχική συζήτηση, δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν, απλά ήθελα να τονίσω την ανάγκη Θα ήθελα να τονίσω τα θέματα που υπάρχουν στην έκθεση αυτή και να τονίσω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στα συστήματά μας να αναπτυχθούν, όχι να περιορίσουμε αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν τους τομείς αυτούς ε, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να εξετάσουν ε, τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ώστε πράγματι να διασφαλίζουν ότι επιφέρουν προστιθέμενη αξία και ότι δεν ε, αντιγράφουν απλά αυτό που μπορεί να γίνει κάλλιστα ε, σε ένα εμπορικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κακόπ. Ε, και εγώ αναφέρομαι συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Φιλανδία. Ε, διότι η κυρία Πάκ ε, ανέφερε ε, ότι κάποιο αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Μπέλετ για το καλό σχέδιο ψηφίσματος του, που το οποίο είναι και ισορροπημένο. ακολουθεί τη γραμμή της ειδικής μου έκθεσης για τον ε, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο. Ε, χαίρομαι λοιπόν που αναφέρει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Κάποιες διευκρινήσεις θα ήθελα. Όσον αφορά το σημείο 9, το θεωρείται αυτό σημαντικό θέμα, συμφωνώ απόλυτα στο, την τελευταία φορά στο Στρασβούργο μπόρεσα να ε, επισκεφτώ το οπτικοακουστικό παρατηρητήριο και κάποιες από τις προτάσεις ε, στην ε, έκθεσή μου έχουν να κάνουν με το ρόλο ε, του Ινστιτούτου αυτού. η διευκρίνηση που θα ήθελα είναι η εξή. Όταν μιλάτε για την εντολή που θα δοθεί στο παρατηρητήριο να παρακολουθούν ε, την κατάσταση στα κράτη-μέλη, το αν τηρούν δηλαδή τα πρότυπα, σε ποια πρότυπα αναφέρεστε. Και θα μπορούσε ίσως κανείς να θεωρήσει ότι το παρατηρητήριο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει και κάποια άλλα καθήκοντα, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα του κρατικού τομέα, ε, των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Αυτό που είπε και ο κύριος Κάκοπ το αν ε, τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα ε, πληρούν τα κριτήρια, αν ε, ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θέλουμε. Επίσης, όσον αφορά το σημείο 40 που αναφέρεστε στους διάφορους ενδιαφερομένους που θα πρέπει να συμμετάσχουν. Η συνεργασία αυτή καθεαυτή ε, γιατί τονίζετε από εσά, ε, ποια είναι η πρόθεσή σα περί τίνο ακριβώ μιλάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κυρία Μπίσκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βοβέλετ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το έγγραφο που έχει υποβάλει αποτελεί πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτησή μας. Έχουν συμπεριληφθεί πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει σε διάφορα επίπεδα στο παρελθόν. Σε κάποια σημεία έχω, κάποια... έχω λίγο πρόβλημα με το παρατηρητήριο οπτικοακουστικών μέσων. Θα πρέπει να ελέγχει περισσότερο τα κράτη-μέλη, να ελέγχει εάν οι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά ε, την ε, κρατική ανεξάρτητη ραδιοτηλεφωνία εάν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές. Εμείς ως Κοινοβούλιο ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα μπορούμε να αναθέσουμε σε παρατηρητήριο να παρακολουθεί τις ε, διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ. Μπερδεύουμε μεταξύ τους διαφορετικά επίπεδα. Θα πρέπει να σκεφτούμε τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα καθήκοντα ενός τέτοιου παρατηρητηρίου. Συμφωνούμε ότι θα είναι χρήσιμο να υπάρχει κάποιο, κάποια ευρωπαϊκή υπηρεσία που να εξετάζει το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και που θα εξετάζει αν οι υποχρεώσεις ε, των ε, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ε, πληρούνται. Αλλά δεν μπορεί να είναι στόχος μας ε, να αναθέσουμε υποχρεώσεις σε υπηρεσίες τη στιγμή που αυτό δεν ε, δικαιολογείται σε πολλά κράτη-μέλη ε, υπάρχει το πρόβλημα με τους κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αφενός ε, της υπερβολικής χρηματοδότησης, αλλά αλλού ε, υπάρχει το πρόβλημα της υπερβολικά χαμηλής χρηματοδότησης. Το βλέπουμε αυτό στην Ισπανία. Χρηματοδοτούνται οι σταθμοί αυτοί από φορολογικά έσοδα φορεί ορίζονται από τα κοινοβούλια των χωρών. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο η, η, πολιτική πλειοψηφία ε, αποφασίζει ε, τη χρηματοδότηση των αντιβλεπτικών σταθμών. Ε, θα πρέπει πράγματι έτσι να γίνεται η χρηματοδότηση. Από την άλλη, αν πούμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να χρηματοδοτείτε σωστά την ε, ραδιοτηλεόραση, τότε δεν μπορεί ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να απειλεί με το ρόπαλο του, της δήλωσης, του νόμου για ε, τις κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ε, κρατική ραδιοτηλεόρασης, ε, κινδυνεύουμε πάντα να συγκρουστούμε με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, αυτό φάνηκε σαφώ πέρσι. Ωστόσο, Υπάρχει απ' την άλλη ο κίνδυνο να διαμαρτυρηθούν ιδιωτικοί σταθμοί και να επιβληθούν κυρώσει σύμφωνα με τον νόμο περί κρατικών ενισχύσεων. Θα ήθελα να πω κάτι στον συνάδελφο Κέρκοπ. Ε, δεν θα ήθελα να μείνει έτσι αυτό που είπε. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίζουν ε, τις υποχρεώσεις της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Τουλάχιστον στη Γερμανία, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη, ε, οι υποχρεώσεις αυτές δεν περιορίζονται σε αυτό που δεν κάνουν οι ιδιωτικοί σταθμοί. Είναι πολύ πιο ευρείες οι υποχρεώσεις. Κοινωνικός ρόλος δεν θα πρέπει λοιπόν απλά να συμπληρώνουν ένα κενό που υπάρχει. Και αναφέρεται αυτό ε, στην έκθεση του Ιβο Πέλετ. Ε, αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο για την πληροφόρηση των ε, πολιτών μιας χώρας. Δεν παίζουν απλά ρόλο κλεισίματος των κενών που υπάρχουν. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα. Το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία είδαμε μια πολύ καλή συνεργασία του κρατικού καναλιού ARD ε, με ε, ιδιωτικό σταθμό το ProSieben. Ε, το προϊόν ήταν η Λένα που κέρδισε τη Eurovision. Υπάρχει ανάγκη και από τις δύο πλευρές για περισσότερη δημιουργικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει συνείδηση και από τις δύο πλευρές. Πολύ συχνά ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο σκληρός όσο συχνά αναφέρεται. θα είναι χρήσιμο να αναθεωρήσουν και οι δύο πλευρές ε, τη θέση τους ε, και είναι χρήσιμο η Ευρώπη να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε να προσπαθήσει να πετύχει την ε, συνάντηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων που είναι σημαντικά για τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ. ich möchte mich auch ο Αντιπρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιβο Μπέλετ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο αυτό. Θα... Μου άρεσε όχι να το υιοθετήσουμε γρήγορα, αλλά να το θεωρήσουμε έγγραφο εργασίας, το οποίο να πρέπει να αναθεωρηθεί, διότι είναι τόσο γρήγορες εξελίξεις στον τομέα της ε, ραδιοτηλεόρασης που βλέπουμε νέες εξελίξεις. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Δεν θέλουμε να υπάρχει χάσμα. Αυτός είναι σημαντικός στόχος. Ωστόσο, όσο καλά και να είναι κάποια ε, ψηφιακά μέσα, τόσο εμβαθύνουν ε, ένα χάσμα που υπάρχει στην κοινωνία μας. Κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα δει κανείς ε, με μια παλιά αναλογική τηλεόραση. 300 σταθμού μπορώ να δω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει τηλεοπτική συσκευή που με ε, μια ειδική κεραία μπορεί να μου προσφέρει 3.000 σταθμού. Αυτό είναι τεράστιο άλμα. Αλλά πολλοί κόσμος ε, δυσκολεύεται να χειριστεί και τις παλιές τηλεόρασεις ε, και οι νέες στοιχίζουν πολλά. Οι αναλύσεις δείχνουν λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ε, ένα σοβερό μειονέκτημα. Όλα εξαρτώνται από τα χρήματα που έχει κανείς στη διάθεσή του. Άλλο είναι να έχει κανείς ε, τηλεόραση που να πιάνει 3.000 σταθμούς και που να επιτρέπει και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ε, η οποία στοιχίζει όμως 3.500 ευρώ. Δεν έχει ο καθένας τόσα χρήματα. Από την άλλη, πολλώνται πολλές ε, συσκευές όπου δεν χρειάζεται ε, επιπλέον ε, όπου δεν ε, χρειάζεται επιπλέον κεραία. Αυτήν συνήθως προτιμάει πολλοί κόσμος στη Γερμανία. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν μια σαφή διαχωριστική γραμμή στην περίπτωση των ανθρώπων που δεν δαπανούν ε, ε, τόσα χρήματα για να αγοράσουν μια τηλεόραση. Ο στόχος λοιπόν ε, της επικοινωνιακής ισότητας είναι πολύ σημαντικός, θα πρέπει να τον τονίσουμε αυτόν. Θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχουν μεγάλες διαφορές, δεν μπορούμε όμως να τις εξαλείψουμε εν μία νυχτή. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρικές αναλύσεις που υπάρχουν. Το άλλο που θέλω να πω έχει να κάνει με την εποπτεία. Έχω προβλήματα με το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος θα αποφασίζει τι θα πρέπει να εξετάζεται. Αντί για παρακολούθηση, θα προτιμούσα ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο στα πλαίσια του οποίου να είναι δυνατή μια ποιοτική εξέταση του αν ε, πληρούνται τα κριτήρια. Υποθέτω ότι αυτό θα ήταν περισσότερο ε, θέμα έρευνας παρά ε, ρόλος ενός παρατηρητηρίου που θα εποπτεύει το περιεχόμενο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να μπορεί να παρέχει πληροφορίες για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ε, τελευταία παρατήρηση είναι μια ερώτηση. Με την ψηφιοποίηση θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής περιφερειακών ε, ή κρατικών προγραμμάτων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Στη Γερμανία είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν ε, ιδιωτικοί σταθμοί, τοπικοί, υπάρχουν δήμοι που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, ε, αλλά όλο και λιγότεροι. Και είναι, είναι δραματική κατάσταση διότι οι μεγάλες πόλεις έχουν τέτοιου τέτοιους ε, ενώ οι μικρές όχι. Οι μικρές πόλεις με ε, λίγους κατοίκους ε, μπορούν να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο μόνο με διαφήμιση. Η διαφήμιση όμως για μία πόλη μόνο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και προσφέρει πολύ λίγα έσοδα. Μήπω θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά την εισαγωγή των ψηφιακών μέσων, να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής ε, ραδιοτηλεόρασης. Ευχαριστώ. Η κυρία Άνιμπαλ. Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι καθόλου σίγουροι ότι έχουμε ένα διπτό σύστημα. Έχουμε παραπάνω από δύο εταίρους. Μιλήσαμε για την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ε, ουσιαστικά γι' αυτό μιλάει αυτή η έκθεση. Και μιλήσαμε για τις, ε, τους εμπορικούς σταθμούς. Αλλά δεν έχουμε διερευνήσει καθόλου το ίντερνετ. την online αναμετάδοση, όλες αυτές τις μορφές αναμετάδοσης που έχουν τεράστια επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο διαδίδονται τα νέα και οι ειδήσει. Ένα από του λόγους για τον οποίο μειώνται οι διαφημίσεις στου εμπορικού σταθμούς, στου ιδιωτικού σταθμούς, είναι ότι οι εταιρείε ε, προτιμούν να διαφημίζουν τα προϊόντα τους online. Βρίσκουμε πάρα πολλές διαφημίσεις ε, στο Google, ε, διαφημίσεις που στο παρελθόν τις βλέπαμε στην τηλεόραση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ρεαλιστική συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα τεκτενόμενα online. Η, ευρωζώνη, η ευρωζωνική κάλυψη βελτιώνεται όλο και περισσότερο ε, και ο κόσμος ε, ενημερώνεται με ένα και διαφορετικούς τρόπους. Ε, πρέπει να γνωρίσουμε τα τεκτενόμενα, τι τεκταίνεται. Εγώ θυμάμαι, κύριε Κιάκο, ε, την εποχή που είχαμε τέσσερα ε, κανάλια. Όλοι παρακολουθούσαμε τα ίδια. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ συνεκτικά. Ε, Πήγαμε στο σχολείο, ας πούμε, και συζητούσαμε τα ίδια προγράμματα. Τα είχαμε δει όλοι. Αυτό δεν ισχύει πια. Δεν υπάρχει αυτό. Πέθανε. Υπάρχει μεγαλύτερος κατακαιρματισμός σήμερα ε, στα ΜΜΕ. Ε, όπως αυτό που είπε ο κύριο Μπίσκι με τον τεράστιο αριθμό των σταθμών και καναλιών. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιο να θέλει πρόσβαση σε παραπάνω από ξέρω, 250 σταθμού. Πάντως η επιλογή είναι ατέρμονη. Και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Πώς αντιλαμβανόμαστε την δημόσια τηλεόραση μέσα σε αυτό το πλαίσιο γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποια ορόσημα, ε, κάποια σημεία αναφοράς. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τον τρόπο που διαδίδονται τα νέα και οι πληροφορίες. Ε, πρέπει να το δούμε όλα αυτά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τι συμβαίνει πραγματικά στην εκπομπή και στους σταθμούς και στην online ενημέρωση. Φυσικά υπάρχει και η γραπτή ενημέρωση που όλο και συρρυκνώνεται με την έλευση του ίντερνετ και την αύξηση της τηλεόρασης και της online αναμετάδοσης. Ο κόσμος έχει όλο και περισσότερες πληροφορίες από όλα αυτά τα μέσα τώρα και νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ε, πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να το δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα συμβαίνουν. Και σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να σκεφτούμε και την ιδιοκτησία των ΜΜΕ. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλοι, τεράστιοι ιδιοκτήτε των ΜΜΕ. Ε, τα μέσα ενημέρωση ε, είναι συγκεντρωμένα σε λίγα χέρια. Και αυτό συνδέεται με τη δημοκρατία και το ζήτημα της δημοκρατίας. Τώρα, για όσα είπαμε για, την, για το παρατηρητήριο, είμαι καθόλου πεπισμένη. Ε, θέλω να ακούσω περισσότερα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό για να πιστώ. Σε αυτή τη φάση δεν μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Δεν νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο στα κράτη-μέλη. Δεν είναι απλώς ε, θέμα Big Brother. Μπορεί να είναι αποδειχθεί απλώς μια τεράστια ευρωπαϊκή αποτυχία και να μην μας βοηθήσει καθόλου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλετ για την έκθεσή του. Ε, είναι μια καλή βάση για μια συζήτηση, για μια ενδελεχή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις παρεμβάσεις. Να επανέλθω αυτό που ο κύριος Μπίσκι Έχουμε διαφορετικά συστήματα. Συστήματα με εισφορά, τέλη δηλαδή, δημόσια συστήματα. Στη Φιλανδία πληρώνουμε ένα τέλος. Αλλά το τέλος αυτό δεν πληρώθηκε από πολλά άτομα. Και το θέμα τότε και όλο το ζήτημα το ξαναείδαμε, το ξανασυζητήσαμε. Διαρωτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να εξελιχθεί το σύστημα. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπέλετ για να απαντήσει. Uh, thanks very much, ε, chairman. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις ακούσαμε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα Ολλανδικά σε κάποιες ερωτήσεις. Σημείο 9. Και την πρόταση να δώσει η Επιτροπή εντολή... Στα Ολλανδικά είπα θα μιλήσω, ζήτω συγγνώμη. Η πρόταση αυτή να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εντολή. Φυσικά δεν θα πρέπει να είναι ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, και να εποπτεύουν ε, τα πάντα. Στόχος δεν είναι ο έλεγχος. Ίσως ο κύριος Πίσκι να πλησίασε περισσότερο αυτό που ήθελα εγώ. Ε, είναι πιο πολύ ε, θέμα έρευνας. Ο κύριος Λούκεκο το ανέφερε αυτό. Έχω επισκεφτεί και εγώ το παρατηρητήριο οπτικοακουστικών μέσων. Είναι πολύ χρήσιμη η δουλειά που κάνουν. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο ε, Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου συμμετέχει στις διαδικασίες. Έτσι μπορούμε να γεφυρώσουμε τις δικές μας υποχρεώσεις από τη μία μεριά και από ε, και τις υποχρεώσεις ε, που επιβάλλει το Συμβούλιο της Ευρώπης από την άλλη διο... Ε, μέσω αυτού του παρατηρητηρίου. Αλλά αυτό που συζητάμε εδώ πέρα δεν είναι μια οριστική έκθεση, είναι μια πρόταση, είναι ένα σχέδιο πρότασης. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στις διάφορες παρατηρήσεις. Ίσως θα πρέπει να πω ότι μία από τις βασικές αιτίε που συνέγραψα την έκθεση αυτή και που ε, ενέκρινε η κυρία Πάκ την απόφαση αυτή ε, στις συνεδρίες των συντονιστών είναι ότι η κατάσταση ε, για είναι η κατάσταση για κάποιες για κάποιους κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ποιο είναι το σημείο κίνησης, δεν μπορούμε όμως να προβλέψουμε απόλυτα το αποτέλεσμα. Εάν σας ε, αναφέρω την κατάσταση στο Βέλγιο θα μου πείτε ότι ναι, αλλά τι γίνεται στο, στην Ουγγαρία ή στην Ιταλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να αποφύγω λοιπόν κάτι τέτοιο. Ελπίζω στην Επιτροπή μας ε, να ε, βρω την κατάλληλη πλατφόρμα εδώ στην Επιτροπή μας. Αν αρχίσουμε απλά να κατηγορούμε έναν στον άλλο δεν θα προχωρήσουμε. Αυτό το έχουμε δει στην Ολομέλεια. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε καλά δομημένες προτάσεις και λύσεις. Σε κάποια κράτη-μέλη διαφέρει η κατάσταση από άλλα κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να υπάρχει υπερβολική χρηματοδότηση των κρατικών ραδιοσταθμών, ε, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ε, σε άλλα κράτη-μέλη όμως ε, μιλάμε για υποχρηματοδότηση και ε, δυσκολεύονται να επιβιώσουν οι κρατικοί ραδιοτηλεοπτικέ σταθμοί. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μήπως θα πρέπει να του βοηθήσουμε λίγο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της νομοθεσίας, ε, της ανταγωνιστικότητας, ε, οι προσφυγές προς την Κομισιόν ενώ σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για το θέμα αυτό. Ο κύριος Πίσκη είπε και τώρα σε άλλο θέμα, ότι υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες με την ψηφιοποίηση. Μπορεί κανείς ε, να ε, λαμβάνει 3.000 σταθμούς ε, στην τηλεόραση, μπορεί να βλέπει περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή στο iPhone. δεν ε, υπάρχει πια το διτό σύστημα. Το διτό σύστημα το έχει καταπιεί ε, το, όλο αυτό το πλαίσιο των μέσων επικοινωνίας. Έχουμε πολύ μέσα. Και γι' αυτό, κύριε Πίσκη, έχετε δίκιο ότι προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει πιο βαθύ το χάσμα αυτό άσχετα από το πού βρίσκεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άσχετα από το κοινωνικό του υπόβαθρο, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των μέσων επικοινωνίας και μάλιστα θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις καλύτερες πληροφορίες ε, στην πιο χαμηλή τιμή. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο αίσθημα ιδιοκτησίας των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, που ανέφερε η κυρία και εδώ τίθεται το θέμα των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο. Όσον αφορά το σημείο 12 του, της πρότασης ψηφίσματος, ε, αναφέρομαι στην διαφάνεια του καθεστώτος ιδιοκτησίας ε, των ε, ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και το θέμα της διασταυρούμενης ιδιοκτησίας. Ε, πάντως υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλετε προτάσεις όπως θέλατε. Και επίσης όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά, αναφέρθηκε το Google και την ε, πίεση που ασκεί το Google στην ε, αγορά της διαφήμισης. Υπάρχουν λιγότερα έσοδα δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, όχι μόνο για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και τα τυπωμένα μέσα που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο δεν ε, έχουν τόσο μεγάλα έσοδα από τις ε, διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Ασκείται σημαντική πίεση από browser όπως είναι ο Google, από μηχανές αναζήτησης όπως είναι το Google, ε, διότι καταπίνουν μεγάλο μέρος των εσόδων. Το γνωρίζουμε αυτό ε, γι' αυτό στην πρότασή μας θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλία, να συζητήσει το θέμα αυτό μαζί μας για να δούμε πώς μπορούμε να υποβάλουμε καλύτερες προτάσεις για το θέμα αυτό. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα της ε, έκθεσης αυτής. Και κύριε Μπίσκη, ναι, σαφώς θα ήταν καλό να καταλάβουν όλοι ότι ε, η λύση αυτή δεν αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που θα πρέπει μάλλον να συγγράφουμε νέα έκθεση κάθε χρόνο για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις του τομέα και για να εξετάζουμε τι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλαμβάνουμε για να ε, ακολουθήσουμε τις εραγνές εξελίξεις σε ψηφιακό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε έτσι τι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε. Σίγουρα δεν έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ή με ε, Βέβαιο όμως ότι στις ε, ε, προσεχείς διμερεί συζητήσει που θα έχω θα λάβω τις σχετικές προτάσεις από τους και Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε την, το σχέδιο έκθεση του κ. Μπελέτ. Είναι πολύ επίκαιρη, ε, πολύ ισορροπημένη αυτή η έκθεση, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποιες αρχικές παρατηρήσεις για το σχέδιο. Καταρχάς, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ε, αναγνωρίζει η έκθεση τη σύσταση της Κομισιόν για τη, το, τις κρατικές ενισχύσεις ε, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ε, οι κανόνες αυτοί δεν έρχεται σε σύγκρουση με το διτό σύστημα, αλλά είναι προϋπόθεση για την ε, ύπαρξη του διτού συστήματος. Είμαστε σε μια φάση όπου οι ιδιωτικοί σταθμοί, οι εμπορικοί σταθμοί δυσκολεύονται πάρα πολύ και είναι σαφές ότι αν δεν υπήρχαν κανόνες για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, ίσως να εξαλειφόταν ε, η εμπορική σταθμή και να μην είχαμε πια διτό σύστημα. Ε, οι κανόνε λοιπόν για τι ε, κρατικέ ενισχύσει, για την κρατική ραδιοτηλεόραση είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα πάντω για το διτό σύστημα. Πολύ κέριο το ερώτημα τη κυρία Χάνιμπαλ. Υπάρχουν πολλές ε, διαφορετικές πλατφόρμες σήμερα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διτό σύστημα. Γιατί Έχουμε κάτι που υποστηρίζεται από την κρατική χρηματοδότηση και από την άλλη έχουμε μια παλέτα από εμπορικέ πρωτοβουλίε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν συζητάμε την αναθεώρηση τη ανακοίνωση με του ενδιαφερομένου, με του stakeholders, μέχρι στιγμή ε, είχαμε πάντα διάλογο μεταξύ των ε, ε, εκπροσώπων της δημόσιας και της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης. Στην τελευταία αναθεώρηση όμως και ο γραπτός τύπος ενεπλάκει πολύ γιατί όλο και περισσότερο υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες στο ίντερνετ και αισθάνονται απειλούμενοι από την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Ε, μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό ε, για τη σημασία του τίτλου συστήματος. Έχουμε το θέμα επίσης της παρακολούθησης, του monitoring. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συνθήκη και ιδίω το πρωτόκολλο για την για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες και τονίζει ότι τα, τα κράτη-μέλη ε, καθορίζουν το εύρος της δημόσιας ε, ραδιοτηλεόρασης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής λέει ότι νέες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πιθανές μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει και χώρος οπωσδήποτε για την επικουρικότητα. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες τώρα για τη δυνατότητα ε, ύπαρξη ή δημιουργία ενός φορέα που θα αποφασίζει ποιο είναι το σωστό επίπεδο δημόσια υπηρεσία. Γιατί τα πράγματα διαφέρουν πολύ από κράτο μέλο σε κράτος μέλος, ε, συνδέεται με κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και κάποια κράτη-μέλη ε, πάντα θα έχουν ένα μικρότερο δημόσιο τομέα από άλλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμοδιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση να του πει ότι δεν είναι σωστό αυτό. Το, για το παρατηρητήριο τώρα. Ε, η φύση του παρατηρητήριου είναι μια μερική ε, συμφωνία που επεκτάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, μερική γιατί δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και είναι εκτεταμένη γιατί συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου συμμετέχουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή στο Παρατηρητήριο. Ε, συμμετέχουμε συζητήσεις μεταξύ όλων των μελών του παρατηρητηρίου για να αποφασίσουμε ποια είναι, ποιες είναι οι και τα καθήκοντα του παρατηρητηρίου. Πρόσφατα έγινε μια συζήτηση για να αυξήσουμε τα καθήκοντα του παρατηρητηρίου για να παρακολουθεί και να εποπτεύει και τις νέες ε, υπηρεσίες. Ε, και η πλειοψηφία των κρατών μελών που πολλά από αυτά δεν είναι και κρατήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν είπαν ναι σε κάτι τέτοιο. Για την πρόσκληση που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμία αντίρρηση. Για το θέμα της διαφάνειας και της ιδιοκτησίας των σταθμών εκπομπής. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με, την, ε, με τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και τελευταία φορά που έγινε μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο δεν υπήρχε πλειοψηφία για να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα. Τώρα, τι έκανε η Κομισιόν. Παραγγείλαμε μια ανεξάρτητη μελέτη για να δημιουργηθούν κάποιοι δείκτες που θα μετράνε την ε, τον πλουραλισμό του ΜΜΕ και να καλυφθεί και το θέμα της ε, διαφάνειας και της ιδιοκτησίας. Υπάρχουν μια σειρά από δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πάντες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για να εξετάσουν την κατάσταση. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προβληματισμού για τις ε, βέλτιστες πρακτικές κτλ. κτλ σας ευχηστώ την προσοχή στην ε, ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν και είμαι σίγουρος ότι η Επίτροπος Κρούς θα σας πει περισσότερα για αυτό το θέμα αύριο. Ένα από τα θέματα που αναφέρει η ψηφιακή ατζέντα είναι η προετοιμασία ε, ενός πράσινου, μιας πράσινης βίβλου για τις προκλήσεις και τις ε, ε δυνατότητες που δημιουργούνται για το δημιουργικό περιεχόμενο. Ευχαριστώ για αυτά τα σημεία. Θα επανέλθουμε στην επόμενη συνεδρία σε αυτό το σημείο, τον Ιούνιο. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε και αυτό το σημείο. Α, είμαστε στην ώρα μας. Δεν έχουμε καθίσει καθόλου. Σαν πραγματικοί Φιλανδοί και Γερμανοί. Ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μουσείων. Πρόκειται για ένα δίκτυο που θα μας το παρουσιάσουν. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους του ΝΕΜΟ στη συνεδρίασή μας. Θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση της Ελιζαμπέτα Πετρούσας Στρούκταν, πρόεδρο του δικτύου, και τον Μάικ Τέιλορ. Δέκα λεπτά ο καθής για τις παρουσιάσεις σας. Εν συνεχεία θα περάσουμε στη συζήτηση. Η κυρία Πέτρουσα Σάστεχαλ έχει το λόγο. Thanks a lot to the... Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή σας για το ότι μπορούμε εμείς ως δίκτυο εκπροσώπων να είμαστε εδώ και να έχουμε τον λόγο για να παρουσιάσουμε στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα θέματα του ΝΕΜΟ. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά χρειάζεται μια ιδιαίτερη δυνατή φωνή υπέρμαχου και για να μπορέσουν μέσω των θεσμικών οργάνων να παρουσιαστεί το έργο μας και να υποστηριχθεί. Η ΝΕΜΟ έχει αυτό το ρόλο να έχει ευδιάκριτο χαρακτήρα που θα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το 1992 ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη ένωση μουσείων και παρόμοια σώματα που εκπροσωπούν την κοινότητα των μουσείων στην Ευρώπη και στις συνδεδεμένες χώρες. Εφέτος, έχουμε κράτη-μέλη από 32 χώρες μέλη. Πολλές από τις ε, οργανώσεις ε, υλοποιούν το έργο τους με μικρή χρηματοοικονομική δυνατότητα και δυναμικό. Πολλή δουλειά την κάνουν οι εθελοντές και μέσα στο πλαίσιο του νέου έχουμε 60.000 ε, ευρώ ετήσια που μπορούν έτσι να χρησιμοποιούνται. Έχουμε μια φωνή επιπλέον όλα τα στοιχεία που αφορούν την ε, πολιτική μας έναντι όσων είναι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής. Θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης. Έχουμε σε τακτά διαστήματα συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητήσεις ε, για όλα τα θέματα που αφορούν τα μουσεία και η ανταλλαγή απόψεων που προωθεί τα θέματα των μουσείων. Ομάδες εργασίας ε, όπως ε, πλατφόρμες ε, και μονάδες για την πρόσβαση στην, στον πολιτισμό, συνεργασία στον πολιτισμικό τομέα και συνεισφορά και input σε διαφορετικά προγράμματα πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, τα, οι αιτήσει συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων, βέλτιστες πρακτικές και θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τα μουσεία και θέσπιση συνεργασίας και επαφών μεταξύ μας. Έτσι έχουμε και ιστοσελίδα και δημοσιεύματα για τη διάχυση των πληροφοριών μας. Έχουμε επίσης ε, τα νεμονιούς και ε, θέματα που αφορούν ενδιαφέροντα των μουσείων μας. Παρέχουμε στοιχεία όσον αφορά τη διάρθρωση, στοιχεία όσον αφορά θέματα που ενδιαφέρουν τη δράση των μουσείων. Έχουμε και νέα προγράμματα και ε, νέες δραστηριότητες. Η ιδέα είναι να υπάρχει μια πλατφόρμα για τους εταίρους για τέτοιου είδους ευρωπαϊκά προγράμματα ή εγχειρήματα. Μία από τις δραστηριότητες μας ε, είναι η δυνατότητα ε, διάδοσης πληροφοριών για συνέδρια, αντίστοιχες επαφές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το νέμο προωθεί και τα μουσεία ως ε, μέσα παιδείας και εκπαίδευσης και έτσι είναι πάροχος υπηρεσιών ε, σχετικά το ναι άρχισε την διάδοση πληροφοριών μέσω της ε, προσπάθειας αυτής διάχυσης των στοιχείων μουσείων όπως και το Ευρωπαϊκά η συλλογή των ειδήσεων και νέων και Ιστοριάνα πληροφορίες για τέτοια θέματα όπως ε, οι προδιαγραφές, η ψηφιοποίηση, ο διαπολιτισμικός διάλογος, ε, δημιουργικότητα και καινοτομία. Βρίσκονται στοιχεία αυτά στις ιστοσελίδες ώστε να μπορούν να μαθαίνουν τα μουσεία το ένα από το άλλο. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Τέιλορ ο οποίος θα σας δώσει κάποια περισσότερα στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. 30.000 λοιπόν μουσεία στην Ευρώπη και υπάρχουν παντού μουσεία που εκπροσωπούν τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών να μπορέσουν να, να τεκμηριώσουν την ιστορία τους και την, το πολιτισμικό τους παρελθόν, να δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσουν οι πολίτες τον περίγυρό τους 500 εκατομμύρια πολίτες επισκέπτονται τα μουσεία αυτά ετήσια. Θέλουμε κάποια από τα θέματα να αναφέρουμε που αφορούν τις δραστηριότητες των μουσείων συνολικά. Όπως είπαμε η κινητικότητα των συλλογών των μουσείων, ο δανεισμός και η εξωτερική παρουσίαση αυτών των στοιχείων μπορούν να δείξουν τις παραδόσεις μας και τις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας η κινητικότητα είναι και έχει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική ατζέντα της ημερήσιας ε, ε, διάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο όσον αφορά διατάξεις για προσωρινές ε, τέτοιες εκθέσεις. Δημοσιεύτηκε το 2007 για να ενθαρρυνθούν οι δανειακές αμφίδρομα αδραστηριότητες, άσχετα από ποιο μέγεθος ή κατηγορία. Και σε 12 ευρωπαϊκές γλώσσες. Ήταν η ιδέα του νέμου, πολύ σημαντική συνεισφορά για την κινητικότητα των συλλογών που θα αποβεί σε μακροπρόθεσμα προς όφελος των πολιτών. Επίσης αποτελούμε <clears throat> τμήμα της κινητικότητας των μουσιακών συλλογών από το Μάη 2007 Περαιτέρω χρηματοδότηση πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διατίθεται για καινοτόμα τέτοια προγράμματα για να καταδειχθεί η πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά στα πολιτισμικά θέματα. Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαία ανταλλαγή στοιχείων για να υπάρχει βαθύτερη κατανόηση των παραδόσεών μα και των ριζών στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε και την, την ομάδα εργασίας OMC για τις συλλογέ μας. Έχουμε πέντε διαφορετικούς τομείς ε, όσον αφορά ε, τις ε, αποζημιώσεις, τις επαγγελματικές επαφές, το μακροπρόθεσμο δανεισμό, το νέμο πιστεύει ότι η κινητικότητα των συλλογών πρέπει να τύχει περαιτέρω προσπάθειας για να μπορέσει να προαχθεί. Αυτό είναι προτεραιότητα σε σχέση με το μέλλον και ενθαρρύνεται η ομάδα εργασίας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με σωστό τρόπο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης για όλες αυτές τις συλλογές που διακινούνται. Τώρα ψηφιοποίηση και ψηφιακή μορφή ιδιαίτερα η νέα γενιά έχει αυτή τη δυνατότητα στο διαδίκτυο να αντλήσει στοιχεία. Πρέπει να είναι λοιπόν προσπελάσιμο αυτό το στοιχείο στο διαδίκτυο. Αυτό ζητείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κληρονομιά αυτή να είναι προσβάσιμος, προσπελάσιμο στους πολίτες μέσω αυτής της πρωτοβουλίας προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα Ευρωπαϊκά έχουν ε, προτεραιότητα και για την ψηφιοποίηση. Είναι γεγονός όμως ότι πολλά μουσεία και ιδιαίτερα μικρά μουσεία βρίσκουν δυσκολίες σε αυτές τις δράσεις. Είναι δουλειά εθνικών ιδρυμάτων ή περιφερειακών ιδρυμάτων να παράσχουν την ε, αρρωγή για την ψηφιοποίηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο πανευρωπαϊκά. Επίσης η υποστήριξη των μικρών μουσείων και για την ψηφιοποίηση των συλλογών τους και η υποστήριξη είναι όπως είπα δύσκολο για πολλά μουσεία να ψηφιοποιήσουν τις συλλογές τους. Έργο του ΝΕΜΟ είναι να ενθαρρύνει αυτές τις προσπάθειες, να υπάρχει κιόλας και ε, ένα φύλλο ενημέρωσης, newsletter για την ψηφιοποίηση και για τα εγχειρήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα Ευρωπαϊκά και το Αθήνα αποκλειστικά θέματα υποστήριξης ευρωπαϊκών μουσείων ώστε να είναι προσπελάσιμα τα στοιχεία στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και η εκπόνηση κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα άλλο θέμα για την ψηφιοποίηση στο διαδίκτυο είναι το θέμα της, ε, του copyright, της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν είναι δυνατόν να, ε, πληρώνουν ε, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των συλλογών τους στο διαδίκτυο. Είναι μη εμπορικά ιδρύματα τα μουσεία δεν έχουν σκοπό την κερδοφορία και έτσι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη αυτός ο χαρακτήρας τους. Παράδειγμα, Ευρωπαϊκά μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνουν αντικείμενα τα οποία είτε δεν καλύπτονται από πλευράς ε, copyright είτε δεν καταβάλλονται τα διότι αυτό μέσα στο πλαίσιο της ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες όταν έχουμε το θέμα της διάθεσης σε ψηφιακό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τη συνεργασία για θέματα copyright από πλευράς μας. Φτάνω τώρα στην παιδεία και εκπαίδευση. Η προσέγγιση της κοινωνίας ε, της μάθησης έχει προτεραιότητα και έχει πολύ μεγάλη σημασία για το έργο των μουσείων πρόσφατα. Πρόσφατα έγγραφα όπως οι δύο ανακοινώσεις του 2009 η πρόοδος ε, για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την παιδεία και την εκπαίδευση και οι αλλαγές μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο ενθαρρύνουν την ιδέα, ενδυναμώνουν την ιδέα ότι η κοινωνική συνοχή, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η αυξημένη προσπελασιμότητα στην πολιτισμική ζωή είναι σημαντικά στοιχεία. Πάλι έχουν κέρια σημασία εδώ και τα μουσεία, όπως η διαβίου μάθηση και εκπαίδευση. Πρέπει να διαδραματίσουμε ένα πιο ζωντανό ενεργό ρόλο στις συζητήσεις η διαβίου εκπαίδευση δίνει μια δυνατότητα στα μουσεία και θέτει νέες προκλήσεις. Είναι ένα φόρουμ έτσι τα μουσεία που συζητώνται θέματα και διασυνδέονται θέματα της διαβίου εκπαίδευσης και μάθησης ώστε να εμπλακούν και να υπάρχει η δυνατότητα προώθησης δυνατοτήτων προγραμμάτων διαβίου εκπαίδευσης για τους πολίτες συνεδριάσεις ε, των εκπαιδευτών ε, και των ε, μελών στην Κοπεχάγη θα διεξαχθεί ένα φόρουμ για να έχουμε και την επετηρίδα της 10ης επαιτίου και έχουμε και την δυνατότητα του δικτύου Γκρούνβικ, το Μουσείο της Μάθησης ή Μάθηση μέσω των μουσείων, υποστήριξη του ΝΕΜΟ ως στοιχείου κλειδιού στην διαβίου παιδεία και εκπαίδευση. Κινητικότητα. Σημαντικό στοιχείο. Πολλά προγράμματα για την κινητικότητα επαγγελματιών μέσα στο πλαίσιο αυτό έχουν συζητηθεί. Δεν έχουμε όμως μέχρι σήμερα ένα πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στα μουσεία. Μέσω ενός τέτοιου προγράμματος οι άλλες πτυχές που ανέφερα μπορούν να ενδυναμωθούν. Ένα νέο τέτοιο πολιτισμικό πρόγραμμα πρέπει να ενθαρρύνει αυτές τις δραστηριότητες, όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά και με κέντρα βάρους μέσα στα ίδια τα προγράμματα. Οι εθνικές υπηρεσίες ε, για τα θέματα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν να ενθαρρυνθούν ε, οι δυνατότητες κινητικότητας των επαγγελματιών στα μουσεία και να δούμε τα κέντρα βάρους στο σχεδιασμό του επόμενου πολιτισμικού προγράμματος. Επίσης, ε, έχει εταίρους το νέμο στις πρακτικές εφαρμογές για την διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιλωτικά για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων, για την ε, φιλική προς τους χρήστες πληροφόρηση, για ε, αλλοδαπούς και εργαζόμενους στον τομέα τον πολιτισμικό που εργάζονται σε κράτη-μέλη. Υποστηρίζει τον ΕΜΟ την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τον ε, Μάρτιο εφέτος για να βελτιωθούν οι δυνατότητες κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών των τεχνών. Επίσης, ε, ο διαπολιτισμικός διάλογος πρέπει να προωθηθεί. Είναι το τέλειο φόρουμ τα μουσεία για να μπορέσει κάτι τέτοια να γίνει κομβικά μέσα στην Ευρώπη και να υπάρξει δυνατότητα επέκτασης ε, μέσω των διαφορετικών εμπλεκομένων. Το ΝΕΜΟ έχει υποστηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες το 2008 είχαμε το έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου με τέτοιες συνέδρια και δημοσιεύσεις και δώσαμε και πληροφοριακά στοιχεία και μέσω του διαδικτύου για τον διαπολιτισμικό διάλογο. After presenting the museum perspective on different... Αφού παρουσιάστηκε η προοπτική ε, των μουσείων, ε, η ΝΕΜΟ θα ήθελε να ε, τονίσει την βασική ανησυχία που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία των μελλοντικών πολιτιστικών προγραμμάτων. Ο ΝΕΜΟ θέλω να αναφερθεί ιδιαίτερα στα μικρά ιδρύματα. Θα πρέπει τα χρηματοδοτικά κανάλια να είναι πιο ευέλικτα για να, υπάρχει, για να υπάρχουν λύσεις για τα μικρά ιδρύματα. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η δομή τους και η, χρηματοδοτική τους, ε, και η οικονομική τους δυνατότητα. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι συνεργασίας με τα μικρά μουσεία, που είναι τα περισσότερα μουσεία στην Ευρώπη και ε, που ε, έχουν την πιο στενή επαφή με τους επισκέπτες τους. Η πολύ ευχαρίστως θα, θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και τους άλλους ευρωπαϊκούς φορείς. και ε, θα καλέσουμε και ε, εθελοντές να συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους της ΝΕΜΟ. Η κυρία Πάκ επέστρεψε, μπορεί να αναλάβει την Προεδρία και πάλι λοιπόν. But I just uh, report and 48 against 5. So I'm, I'm very happy. 48 υπέρ, 5 ε, κατά. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένη. Ήθελα απλά να σας πω 96 ε, τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι ήταν σημαντικό επίτευγμα. πάση, Σας ευχαριστώ όλου. Ε, κλείνουμε λοιπόν τώρα την ε, δημόσια συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε τώρα με την... Ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ όποιος δεν είναι συντονιστής ή βοηθός συντονιστού να αποχωρήσει από την αίθουσα. No, did you, I understand that you No, I just said that it... Ah, you Okay, so I, I Ζητώ συγγνώμη. Παρεξήγησα τελείως την κατάσταση, αλλά φαντάζεστε. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Ποιος ήθελε λοιπόν ε, να ε, θέσει ερωτήσεις. Please. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, καθότι προέρχομαι από μια πολύ μικρή ε, ομοσπονδία της Σλοβενίας, μια πολύ μικρή, ε, ένα πολύ μικρό φορέα. Ε, άκουσα για τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο. Μερικές φορές κάθομαι μπροστά στη τηλεόραση, βλέπω ποδόσφαιρο και αναρωτιέμαι τι θα πρέπει να γίνει με τα μουσεία, ώστε ο κόσμος αυτός να έρθει να επισκεφτεί ένα μουσείο. Πολλοί κόσμος επισκέφτεται τα μουσεία. Αλλά μπορώ να κάνω και την εξής παρατήρηση. Πολλοί κόσμος έχει φύγει τώρα, αλλά η πολλοί κόσμος αποχώρησε, αλλά ε, εσείς που παραμείνατε εδώ πέρα γνωρίζετε το πρόβλημα του έφραυστου τομέα μας. Ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα είναι η παράδοσή μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά. Αν χαθεί, αυτό θα είναι μη αντιστρέψιμο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που βρίσκεστε ακόμα εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Πάκ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, διότι μόλις ε, θυμήθηκα ότι είχα μια συνάντηση με το ΝΕΜΟ πριν 1,5-2 ε, χρόνια. Άκουσα τα ίδια πράγματα, αυτά που μας είπατε σήμερα με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού του Κοινοβουλίου επισκεφτήκαμε τη Στοκχόλμη, όπου προσπαθήσαμε να επισκεφτούμε ένα τέτοιο μουσείο και ήταν εξαιρετικό. Δεν θα το είχα επισκεφτεί αν δεν είχα ενημερωθεί από τους ανθρώπους αυτούς. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να διαδώσετε περισσότερο τις πληροφορίες αυτές ε, στις εκλογικές μας περιφέρειες όταν ε, λοιπόν ε, ο κόσμος επισκέπτεται ένα μέρος, να μην επισκέπτεται μόνο τα σύγχρονα ε, μουσεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά να επισκέπτεται και τα μουσεία που δίνουν μια εικόνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της παράδοσής μας. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Σμιτ, παρακαλώ. Να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ναι, ίσως ε, να οργανώσετε αγώνες ποδοσφαίρου στα μουσεία. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν τομέα που έχω δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα, τον, την εκπαίδευση στον τομέα του πολιτισμού. Είσαστε ένα δίκτυο μεταξύ των μουσείων. Και αν κατάλαβα καλά, ε, ακούγοντάς σας και διαβάζοντας το έγγραφο, προσπαθείτε να φέρετε σε επαφή μεταξύ τους τα μουσεία και να προωθήσετε δράσεις περί ανταλλαγή καλών πρακτικών κτλ. Στις δράσεις σας προβλέπετε κάτι για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Εγώ στη Γαλλία έχω δουλέψει ε, σε ένα τομέα στην Νότια Γαλλία προσπαθώντας να προωθήσω της, την διαπαιδαγωγική διάσταση των μουσείων. Ε, επισκέφτηκα τις, ε, ένα μουσείο στη Στοκχόλμη με την Τόρις. Ε, υπάρχουν τέτοιες ε, παιδαγωγικές δράσεις για τα παιδιά θερυπινική. Ξεκινώντας από τα παιδιά και μόνο αν τα, τους δώσουμε κίνητρα για να επισκέπτονται από νωρίς τα μουσεία ε, θα έρχονται και ενήλικες. Στο πρόγραμμα Grundvig το πρόγραμμα μαθητείας Grundfig, υπάρχει μία δραστηριότητα μεταξύ διαφόρων οργανώσεων για την ε, α, διαπαιδαγώγηση των ενηλίκων, ακριβώς για τα μουσεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδέες στις οργανώσεις των ενηλίκων για να προσαρμοστούν ε, ε, και να συλλάβουν τις άπειρες δυνατότητες που υπάρχουν. Ε, εγώ δεν γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η ιστορία με τα μουσεία. Χάρη ε, στον Νέμο γνώρισα αυτό το δίκτυο. Θα συνεχίσω να μιλάω για αυτό, τον, για αυτό το δίκτυο δεξιά και αριστερά και νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να διαδώσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την, αυτές τις γνώσεις. Πώς είμαστε εδώ πέρα, 8 άτομα. Ε, κάτι είναι αυτό αν ε, μιλήσει ο καθένα από του 8, θα μας ακούσουν πολύ περισσότεροι. Υπάρχει κανένα άλλος που θέλει να παρέμβει. Όχι. Ευχαριστώ τους δύο ε, εκπροσώπους ε, του ΝΕΜΟ που αναγκάστηκαν να, μιλ... να ακούσουν όλα όσα υπόθηκαν για το ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, το ποδόσφαιρο ενδιαφέρει τα πλήθη. Εμείς εκλεγόμαστε από τους ε, ψηφοφόρους μας και με τη σειρά μας θα πρέπει να τους ευαισθητοποιήσουμε για τη σημασία των μουσείων. Λοιπόν, τώρα κλείνω αυτή τη συνεδρίαση και πάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Είναι κανείς εδώ? Μία Τέσσερις.